Καλώς ορίσατε. Η σημερινή δημόσια ακρόαση εγκρίθηκε από το Διευρυμένο Προεδρείο στις 27 Σεπτεμβρίου του 2011. Τρεις ειδήμονες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην ακρόαση αυτή. Επίσης πρόσκληση εστάλει στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καταρχάς θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τους ειδήμονες ομιλητές της παρούσας ακρόασης και να τους ευχαριστήσουμε για τη συμβολή τους εξ ονόματος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Τον κύριο Εμμανουέλ Τζακόπ, πρόεδρο της Euromil, Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Στρατιωτικών Σύνδεσμων, οργανισμό που αντιπροσωπεύει το ευρύ φάσμα των στρατιωτικών οργανώσεων στην Ευρώπη, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τον κύριον Μπένχαρτ Γκέρτζ, επίτιμο πρόεδρο του Σωματείου των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τον κύριο Εμίλιο Αμιράλια, που προεδρεύει το Ιταλικό Σωματείο για την Αλληλεγγύη, τα δικαιώματα και την πρόοδο. Το δικαίωμα του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ήδη από το βασικό κείμενο της Διεθνούς Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτή τη βάση, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ειδικευμένο οργανισμός του ΟΗΕ, επιβεβαίωσε ήδη από το 1919 την αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθε ως μέσο για την βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθεαυτή καθώς και τα κράτη-μέλη της έχουν προσχωρήσει σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό, όπως άλλωστε και κάθε δικαίωμα, υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς και αυτό προβλέπεται ρητά και στις διεθνείς συμβάσεις. Τα κράτη έχουν την δυνατότητα να περιορίζουν τη χρήση του δικαιώματος αυτού μεταξύ άλλων και στις ένοπλες δυνάμεις. Έτσι μερικά κράτη όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι στους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ενώ άλλα κράτη όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Δανία, η Φιλανδία, η Ουγγαρία το αναγνωρίζουν. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει κάποια εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο θέμα αυτό εάν θέλουμε να δημιουργηθεί στο μέλλον μια πιο στέρεη βάση στις κοινέ στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις και αποστολές. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νοέμβρη του 2008 αποτελεί καθαρή ένδειξη προς την κατεύθυνση αυτή. start our discussion today. Θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Εμμανουέλ Ζακόμπ, πρόεδρο της Euromil. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όπως ήδη Είπατε ε, πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία στην εισαγωγή σας, όχι για μένα, αλλά για το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα. Η Υποεπιτροπή ε, για, την, ε, και για την άμυνα και την ασφάλεια ε, θα συζητήσει σήμερα το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε στις ε, ένοπλες ε, δυνάμεις. Ξέρω ότι οι περισσότεροι που συμμετέχονται γνωρίζουν τη Euromil ως σύνδεσμο, ως ένωση, αλλά θέλω να πω και εγώ λίγα λόγια για την μορφή, τη φύση της Euromil. Μετά θα αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία για το δικαίωμα του συνέρχεστε ή συνεταιρίζεστε ε, από στις ένοπλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα αναφέρω ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα. Η Euromil είναι μια ε, οργάνωση γενική, η οποία καλύπτει πάρα πολλούς συνδέσμους και ενώσεις. Ιδρύθηκε το 1972, περίπου 42 χρόνια 40 ε, χρόνια λειτουργεί, έχει 42 ε, συνδεδεμένες ε, ενώσεις ε, από 27 χώρες, εκ των οποίων 24 είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου μισό εκατομμύριο ε, μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών του είναι μέλη και επίσης έχει διαπίστευση και αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ΔΑΣΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και επίσης συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εάν τώρα δείτε το χάρτη της Ευρώπης, οι χώρες με κίτρινο χρώμα είναι οι χώρες όπου η Euromil έχει σήμερα συνδεδεμένες ενώσεις ενώσεις μέλη δηλαδή, συνδέσμους μέλη. Είναι, όπως σας είπα, 27 ευρωπαϊκές χώρες, 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχουν ακόμα ορισμένες χώρες με κόκκινο χρώμα. Είναι χώρες που δεν είναι πλήρη μέλη της Euromil, αλλά έχουν καθεστώς παρατηρητού που σημαίνει ότι έχουν ε, ενεξελίξει έναν σύνδεσμο, ε, αναπτύσσεται δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα σύνδεσμος, ε, των μια στρατιωτική ένωση, ένα στρατιωτικό σύνδεσμο σε αυτές τις χώρες που αργότερα μάλλον θα γίνει πλήρες μέλος. Εν συνεχεία, οι χώρες με γκρι χρώμα δεν εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή στη Euromol, που δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία οργάνωση ή ένωση ε, στις ένοπλες δυνάμεις, ε, αλλά οι οργανώσεις ή οι σύνδεσμοι που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες δεν είναι μέλη της Euromil. Επίσης, στις γκρι ε, χώρες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις στρατιωτικές. Η Αστρία, παραδείγματο υπάρχει συνδικαλισμός στις ένοπλες δυνάμεις, το ίδιο και στην Ορβηγία αλλά όπως σας είπα οι χώρες που είναι σκιασμένες με γκρι δεν είναι μέλη της Euromil. Η αποστολή της Euromil είναι να εκπροσωπεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα επαγγελματικά συμφέροντα των ενόπλων δυνάμεων να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και ζωής, να παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας και την, το σεβασμό και την εφαρμογή των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρώπης, της άνοπλης δυνάμεις. Όταν μιλάμε για το δικαίωμα του δεν εννοούμε ότι ε, κάθε μέλος έχει την δυνατότητα και την ελευθερία να οργανωθεί μέσα στο πλαίσιο των θεμελιωδών ε, πολιτικών δικαιωμάτων που ισχύουν και καλύπτουν όλους τους πολίτες. Ε, αυτό το δικαίωμα του Συνεταιρίζεται λοιπόν είναι ένα από τις πιο σημαντικές αρχές, τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα της Euromil. Διότι είμαστε πεπισμένοι ότι αν η Euromil θέλει να συνεχίσει να είναι ο οργανισμός που ομιλεί εκ μέρους των Ευρωπαίων στρατιωτών, ε, και των μελών των ενόπλων δυνάμων πρέπει ακριβώς να σέβεται και να παρακολουθεί την σωστή εφαρμογή όλων των ανθρωπίνων και σεμελιωδών δικαιωμάτων και του τελευταίου στρατιώτη στις ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης. Το δικαίωμα του συνεστερίζεστε τώρα. Ε, πάντοτε αναφερόμαστε στο δικαίωμα αυτό με διάφορες ερμηνείες από διεθνή κείμενα και συμβάσεις και χάρτες. Οι διεθνείς αυτές συμβάσεις και χάρτες αποτελούν τη βάση της οργάνωσής μας ε, για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Όχι μόνο για το ιδιωτικό προσωπικό, αλλά και όμως δείτε το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες. Διότι το άρθρο αυτό, το άρθρο 11 λέει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελεύθερης και ειρηνικής ε, συμμετοχής σε ενώσεις και συνδέσμους με άλλους ε, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος δημιουργίας και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης, αν δείτε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, άρθρο 5, και πάλι ομιλεί για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε για εργαζόμενους και εργοδότες και ο θεμελιώδης χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρθρο 12 λέει ότι και πάλι όλοι οι πολίτες καλύπτονται και δικαιούνται το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε ε, με ειρηνικό τρόπο και την ελευθερία του συνεταιρίζεστε σε όλα τα επίπεδα τα θεμελιώδη δικαιώματα τώρα του θετικού προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Κοινοβούλιο. Ήδη το 1984 εκδόθηκε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο ζητούσε την αναγνώριση του δικαιώματος του συνεταιρίζοντα στα μέλη των ε, ενόπλων δυνάμεων. Λέει λοιπόν το ψήφισμα του 1984 ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσφέρουν το δικαίωμα σε όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να εδραιώσουν τις ε, επαγγελματικές συνδικαλιστικές τους οργανώσεις και να συμμετέχουν σε αυτές. Το 1995 επίσης εκδόθηκε μια ετήσια έκθεση με τίτλο «Παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» και το άρθρο, η έκθεση αυτή αναφερόταν στο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Um, the European Parliament... Σε αυτή την έκθεση, παραδείγματο χάρη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί και πάλι τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν κανονισμούς για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε στις ένοπλες δυνάμεις και για τους τελούντες, εκτελούντες τη θητεία τους, αλλά και για τα μόνιμα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Το 95 τα δικαιώματα αυτά, ιδιαίτερα για τους υπηρετούντες τη θητεία τους, ε, δικαιολόγησε, καθιέρωσε το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε. Επίσης ε, υπάρχει και η σε θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004-2008. Βλέπω ότι λείπει το 8 από το, ε, την διαφάνεια. Λοιπόν, 2004-2008 ε, ε, αναφέρει λοιπόν ε, η έκθεση αυτή ότι τα σεμελιώδη ε, δικαιώματα ορίζουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους στρατιωτικούς δεν σταματούν στην είσοδο των στρατοπέδων αλλά εφαρμόζονται απόλυτα και σε όλους τους πολίτες, τους ένστολους πολίτες και συστήνει στα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων αυτών και θεμελιωδών δικαιωμάτων στις ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, στο επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει γίνει πολλή δουλειά ε, προς την ίδια κατεύθυνση. Το 1988 ψηφίστηκε το ψήφισμα 903 για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Το 2002 ε, επίσης εκδόθηκε μία σύσταση για την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και το 2006 ανανεώθηκε ε, η σύσταση αυτή με αριθμό 1742. Ε, εν συνεχεία καταφέραμε να εκδώσουμε μία σύσταση από το, την Επιτροπή Υπου, την, Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκε στις 24 Δευτέρου 2010 από τους αναπληρωτές υπουργούς ε, και αναφερόταν ακριβώς στο δικαίωμα του τερίζεστε Και το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε ένα ολοκληρωμένο κείμενο το οποίο έχει εκδώσει σε ένα μικρό βιβλίο οδηγό σε μικρό εγχειρίδιο το οποίο αναφέρει όλες τις συστάσεις και λέει ακριβώς αυτή η σύσταση ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί σε μία περίοδο δύο ετών, άρα το 2012 θα γίνει μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση και επανεκτίμηση αυτής ε, της σύστασης στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Προχωρώντας τώρα στην ΔΑΣΕ, η οποία και αυτή αναφέρεται στα θεμελιώδη δικαιώματα στρατιωτικού ε, προσωπικού, Παραδείγματο χάρη αναφέρεται στο καταστατικό λειτουργίας, στην, ε, στον κώδικα δεοντολογίας, ε, στα θεμελιώδη δικαιώματα. Βλέπετε λοιπόν κυρίες και κύριοι μία εντελεχή τεκμηρίωση που αναφέρεται συγκεκριμένα σε στοχιωτικό προσωπικό και στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ε, και αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα δικαιώματα. Όμως ε, στο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής ε, Σύμβασης υπάρχει και ένα διατάφτα ή ένα όμως, ένα, μια αντιθετική άποψη και λέει ότι ε, καμία ε, αντίθεση δεν θα πρέπει να προβληθεί στην εξάσκηση αυτών των δικαιωμάτων παρά μόνον εάν τίθεται πρόβλημα εθνικής ασφάλειας και ασφάλειας του κοινού και δημόσιας ασφάλειας για την πρόληψη αναταραχών ή εγκληματικών ενεργειών για την προστασία της υγείας και του ήθους και την προστασία των δικαιωμάτων και της ελευθερίας των άλλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι έχει καθιερωθεί, έχει εδρεωθεί και προστατεύεται, όμως μόνο εάν υπάρχουν ειδικές, ειδικά προβλήματα τα οποία ε, αναφέρονται σε θέματα εθνικής και δημόσιας ασφάλειας μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό το δικαίωμα. Επίσης υπάρχουν πολλές ε, ε, αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς ε, την ίδια κατεύθυνση. Αναφέρομαι σε μία περίπτωση του 2008 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε, στην περίπτωση Ντεμίρ, και Μπαϊκάρα εναντίον Τουρκίας όπου τα δύο αυτά, οι δύο αυτοί οι συνδικαλιστές που δεν ήταν στρατιωτικοί είχαν πρόβλημα με την τοπική, τους, ε, με την τοπική αυτοδίκηση, με την τοπική κυβέρνηση για τις λογικές διαπραγματεύσεις. Και ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπε ότι ε, τίθεται, είναι αναγκαία ο σεβασμός των δικαιωμάτων αλλά Επίσης, ενδέχεται ε, να τεθούν ορισμένοι περιορισμοί στις άνοπλες δυνάμεις στην αστυνομία και σε, άλλες, ε, σε άλλα όργανα δημόσιας τάξης. Όμως ε, αυτά, αυτές οι περιορισμοί δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την ουσία του δικαιώματος συνεταιρίζεστε. Ε, και ότι οι εθνικές κυβερνήσει πρέπει να δείχνουν ότι υπάρχουν πιεστικοί λόγοι για τον περιορισμό αυτών των δικαιωμάτων. Μπορούν λοιπόν να υπάρχουν περιορισμοί, αλλά σε πολύ περιορισμένε περιπτώσεις και μόνο όταν υπάρχει απόλυτη και σαφή δικαιολογία. Τώρα, μετά από αυτή την σύντομη ανασκόπηση πρέπει να δούμε τον ρόλο των στρατιωτών. Ο ρόλος ε, των στρατιωτών, ε, του στρατού γενικά έχει αλλάξει. Δεν είναι ο ίδιος ε, στρατός με την ίδια φύση, αν θέλετε, του περασμένου αιώνα. Ο, ο στρατιωτικός, ο στρατιώτης είναι κάποιο, είναι ένα άτομο ένστολο το οποίο συμμετέχει σε διάφορες εκστρατείες. Παραδείγματο χάρη, ειρηνευτικές, μη πολεμικές και έτσι ο στρατιώτης σήμερα γενικά ε, δεν είναι μόνο πολεμιστής, αλλά είναι και ένας διαμεσολαβητής. Είναι ένας διάμεσος ε, ο οποίος ε, ενεργεί για την διασφάλιση των θεμελιών δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Είναι λοιπόν αδιανόητο και αδικαιολόγητο, θα έλεγα και παράλογο, να βλέπουμε στρατιώτες να υπερασπίζονται τα δικαιώματα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του συνεταιρίζεστε σε άλλες χώρες για άλλους πολίτες και να μην μπορούν οι ίδιοι να χαίρονται αυτών των δικαιωμάτων. Να χαίρουν, συγγνώμη, αυτών των δικαιωμάτων. Όπως σας είπα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, επιτυχείς ε, τέτοιες, ε, επιτυχημένες ενώσεις στην Αυστρία, στη Ιρλανδία, στο Βέλιο κλπ. Αλλά σε άλλες χώρες όπου δεν υπάρχουν τέτοιες ε, οργανώσεις, τέτοιοι σύνδεσμοι και άλλες χώρες όπου αυτοί οι κανόνες δεν εφαρμόζονται καθόλου. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες όλων των ευρωπαϊκών χαρών, αλλά αν δείτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι συμβαίνει, γεωγραφικό επίπεδο, οι χώρες σε κίτρινο χρώμα έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα Εκεί υπάρχουν. Όσε χώρε είναι με πράσινα, εκεί υπάρχουν τα δικαιώματα του συνεταιρίζεστε πολλέ φορέ λίαν περιορισμένα και οι χώρες με κόκκινο δεν έχουν τίποτα. Ούτε συνδικαλιστικά δικαιώματα, ούτε δικαιώματα του συνεταιρίζεστε. Και αν δείτε στη Βόρεια Ευρώπη και στην Κεντρική την κατάσταση που επικρατεί, θα δείτε ότι εκεί υπάρχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και είναι πολύ περίεργο να βλέπουμε ότι στα Βαλκάνια και στη Νότια Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα απολύτως. Ακόμα και αν δείτε τον χάρτη αυτόν, ε, θα διαπιστώσετε ότι προσπαθούμε να δείξουμε μία αισιόδοξη εικόνα, ε, διότι χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία, εκεί ισχύει το δικαίωμα του τερίζεστε, αλλά ε, το δικαίωμα αυτό δεν συνεπάγεται και πραγματικά δικαιώματα για τους στρατιώτες. Οι οργανώσεις αυτές που επιτρέπουν το δικαίωμα τους συνεταιρίζεσαι είναι, συν, είναι συνήθως οργανώσεις αποστράτων ή επίτιμων μελών. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην ε, ε, προστασία και βοήθεια στρατιωτικού προσωπικού και μια ειδική περίπτωση είναι της Πορτογαλίας όπου σε κάποια περίπτωση νομίζω το 2001-2002 η πρωτοβολία αποφάσισε να δώσει το δικαίωμα του να σε θετικούς, αλλά ε, επί χρόνια και χρόνια δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί το δικαίωμα αυτό. Και αυτό δημιουργεί εντάσεις, εντάσεις. Η Ισπανία επίσης είναι με πράσινο χρώμα που σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα συνεταιρίζεστε, αλλά είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Μέχρι πριν από δύο μήνες ε, οι στρατιωτικοί δεν είχαν απολύτως κανένα δικαίωμα. Τώρα η κατάσταση άλλαξε, οι ισπανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, όχι το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε. Θέλω να τονίσω ότι πριν από τρία χρόνια στην Ισπανία είχαμε τον πρόεδρο μιας στρατιωτικής ένωσης, ενός στρατιωτικού συνδέσμου που πήγε στη, στη φυλακή δύο φορές επί 30 μέρες, διότι μίλησε δημόσια για το δικαίωμα αυτό. Έτσι, όμως, μέσα σε τρία χρόνια καταφέραμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση στην Ισπανία και τώρα υπάρχει αυτό το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δείτε γενικά, υπάρχει μια θετική εικόνα για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε αλλά όμως ακόμα 11 χώρες δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Μόνο 8 χώρες έχουν το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε με συλλογικές διαπραγματεύσεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν εν κατακλείδη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα για το στρατιωτικό προσωπικό είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ευρώπη. Το, το δικαίωμα του συναστερίζεστε για στο προσωπικό δεν υπονομεύει σε καμία περίπτωση τη στρατιωτική εξουσία ε, και την αλυσίδα ιεραρχίας. Επίσης δεν ε, διακυβεύει την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων και την πειθαρχία εντός των ενόπλων δυνάμεων όταν δίνεται δικαίωμα συνεταιρίζεστε στους στρατιώτες. Δεν διακυβεύεται λοιπόν κανένα δικαίωμα ούτε η ιεραρχία ούτε η πειθαρχία. Πολλές φορές το επιχείρημα που οκογόταν στο παρελθόν ήταν ότι το δικαίωμα αυτό του συνεταιρίζεται θα αποτελούσε ένα μεγάλο πρόβλημα ή θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα. Αλλά μετά από ενδελεχή έρευνα και ανάλυση που έγινε διαπιστώσαμε ότι κανένα πρόβλημα δεν ε, δημιουργείται. Για παραδείγματο χάρη, αν δείτε την Φιλανδία, κανένα δεν μπορεί να πει ότι οι ένοπλε δυνάμει του δεν λειτουργούν εξαιρετικά καλά. Άρα λοιπόν δεν τίθεται κανένα ζήτημα αποδυνάμωσης ή υπονόμευσης της αισθητιωτικής επάρκειας. Το θέμα είναι ότι δεν μας αφορούν οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες και πώς θα αποκαλέσουμε αυτές, αυτά τα δικαιώματα, αλλά πώς θα τα ε, εφαρμόσουμε και τι ουσία θα περιέχουν. Το περιεχόμενο μας ενδιαφέρει, όχι οι τίτλοι. Πρέπει λοιπόν κάποιος να υπεραμείνεται και να υπερασπίζεται αυτά τα δικαιώματα και να μην φοβάται. Ε, μερικές να μιλήσει, να μην φοβάται να μιλήσει. Μερικές φορές, παραδείγματο χάρη στη Γαλλία, ε, υπάρχει μια γενική επιφύλαξη, θα έλεγα μια γενική φοβία να χρησιμοποιηθεί ο όρος συνδικαλισμός, συνδικαλιστής, συνδικαλίζεστε. Ε, όμως είναι γεγονός ότι οι στρατιωτικοί, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνονται για να μπορούν να υπερασπίζουν το επάγγελμά τους και τα δικαιώματά τους. Ε, στην Γαλλία, παραδείγματος χάρη, στην, στο Ενωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία, αυτά τα δικαιώματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγιναν προσπάθειες να οργανωθούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο ή προσπάθησαν τέλος πάντων να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Αλλά τίποτα δεν έγινε, που σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφερόντουσαν καθόλου για τέτοιες κινήσεις. Όμως, όπως είπαμε, ένας στρατιώτης είναι ένας ένστολος πολίτης. Ε, άρα, λοιπόν, Άρα λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι όταν χυθεί το αίμα ενός στρατιώτη είναι το ίδιο κόκκινο όπως το αίμα ενός πολίτη. Άρα λοιπόν, εφόσον το ίδιο αίμα χύνεται και έχει και το ίδιο χρώμα, τα ίδια δικαιώματα πρέπει να ισχύουν και για τους πολίτες και για τους στρατιώτες. Ε, και επίσης πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα του περιορισμού των δικαιωμάτων. Άλλο περιορισμός των δικαιωμάτων σε έκτακτες καταστάσεις και άλλο μηδενική ε, ανοχή στα δικαιώματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν υπεραμείνεται και υπερασπίζεται αυτά τα δικαιώματα και πρέπει θερμά να ευχαριστήσουμε ρωτήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υπεράσπιση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε για τις εκατοντάδες χιλιάδες ε, των στρατιωτικών, ε, των μελών των ενόπλων δυνάμεων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή σχόλια. Σας ευχαριστώ κύριε Τζέικομπ. Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Μπέρναρντ Γκέρτς από την γερμανική, ε, από το γερμανικό ομοσπονδιακό στρατό, την Bundeswehr. Ένωση σωματείων του, της Bundeswehr. the next slide doing this. Okay, thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχω επιφορτιστεί σήμερα με το καθήκον να σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση, μία σύνοψη, αν θέλετε, του γερμανικού προτύπου χορήγηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε για το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ας αρχίσω με τη νομική βάση, το γερμανικό σύνταγμα, στο άρθρο 9 παράγραφος 3 χορηγεί σε κάθε πολίτη το δικαίωμα να προσχωρεί σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επαγγελματικές ενώσεις. Coalition τη γερμανιστή. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε για το στρατιωτικό προσωπικό, ούτε για τις αστυνομικέ δυνάμεις, δεν προβλέπονται δηλαδή στη γερμανική νομοθεσία. Εάν ε, επρόκειτο να υπάρξουν περιορισμοί, έπρεπε να αναφερθούν σε αυτό το σύνταγμα βασική αρχή της θέσης ε, των Γερμανών στρατιωτών ε, μέσα στην κοινωνία είναι η ιδέα του ένστολου ε, πολίτη. το προβλέπεται στο άρθρο 6 του νόμου περί στρατιωτικού προσωπικού και παραθέτω από αυτόν τον νόμο κάθε στρατιώτης έχει τα ίδια δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα όπως και οποιοδήποτε άλλος πολίτης. Σχετικά τώρα με την ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος για την εκπροσώπηση των επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις ενόπλες δυνάμεις. Ε, στις 14 Ιουλίου του 1956, ένα χρόνο μετά την έναρξη δηλαδή του επανεξοπλισμού της Γερμανίας, ε, η Ένωση των Γερμανικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ιδρύθηκε ε, ιδρύθηκε ως επαγγελματική ένωση, σωματείο και όχι ως συνδικαλιστική οργάνωση. Και ο λόγος είναι ότι τότε, τη δεκαετία του 50, το γερμανικό συνδικαλιστικό κίνημα ήταν άρδιν κατά του ε, επανεξοπλισμού. Οπότε... Όταν θέλετε, εφόσον υπηρετεί σε ένοπλε δυνάμει να εκπροσωπηθείτε, αλλά οι συνδικαλιστικέ οργανώσει είναι κατά, αναγκάζεστε να ιδρύσετε μια επαγγελματική ένωση. Σήμερα τα μέλη ανέρχονται σε 200.000, είναι φυσικά σε εθελοντική βάση, είναι ανεξάρτητη ένωση ε, από την κυβέρνηση και από τα πολιτικά κόμματα. Τα, οι δε δαπάνε καλύπτονται από τα τέλη που καταβάλουν τα μέλη και δεν υπάρχει καμία απολύτω επιχορήγηση από την κυβέρνηση. Οι επαγγελματικέ ενώσει και οι συνδικαλιστικέ οργανώσεις στις γερμανικέ ένοπλες δυνάμει, έχουν ειδικά δικαιώματα. Θα προβλέπονται διαβουλεύσει κατά την προετοιμασία των γενικών κανονισμών ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση των στρατιωτών. Αυτά προβλέπονται στο νόμο περί στρατιωτικής υπηρεσίας, στρατιωτικού προσωπικού μάλλον, άρθρο 35α. Όταν ο Υπουργός, ο Υπουργός Άμυνας ε, καταθέτει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, προβλέπεται να μοιράζεται το νομοσχέδιο ούτω ώστε να διαπιστώνετε τι προβλέπεται σε σχέση με τις ε, επαγγελματικέ ενώσεις ε, μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ε, αν έχετε το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και ιδρύζετε μια τέτοια ένωση, όπως σε κάποιες ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν υπάρχει ρύθμιση για την ε, προσχώρηση των μελών, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε εμεί αυτήν την πρόνοια. Ε, μπορεί, μπορούν οι ενώσεις να προσιλητίζουν, αν θέλετε, ή να βρίσκουν νέα μέλη ε, την ώρα υπηρεσίας, ακόμη και στο στρατόπεδο. Ε, δικαιούνται επίσης να συνέρχονται επιτόπου στους στρατώνες ε, εν ώρα υπηρεσίας, αλλά χρειάζονται πρώτερη άδεια του διοικητή. Επίσης, ε, ζητείται από τους διοικητές να επικουρούν τις ενώσεις όπου χρειάζεται μετά από έγκριση του Υπουργού Αμήνης. Υπάρχουν επιπρόσθετες ρυθμίσεις που δεν προβλέπονται στην νομοθεσία αλλά σε συμβάσεις. Ο Σύλλογος των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων έχει συγκεκριμένα σύμβαση με το Γερμανικό Υπουργείο Αμήνης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Το περιεχόμενο έκειται βασικά στην πρόβλεψη ότι δισετησίως τουλάχιστον συνέρχεται ο Υπουργός με τον Πρόεδρο της Ένωσης για μια επίσημη συζήτηση Επίσης, ε, ε, η διοικητικό προσωπικό των δύο αυτών Υπουργείων και οι εκπρόσωποι των ενώσεων ε, συσκέπτονται επίσης προετοιμάζοντας τα νομοσχέδια, ούτω ώστε να μπορέσει να προσφέρει τεχνογνωσία και να ασκήσει επιρροή η Ένωση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όταν εκπονείται κάποιο νέο νομοσχέδιο. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται μέσα στο σχέδιο πρέπει να συζητηθεί ε, σε άμεση επαφή του εκπροσώπου ε, της Ένωσης και ενός υφυπουργού, παραδείγματος χαρές. Περάσουμε στην άσκηση πίεσης. Ε, το γνωστό lobbying. Η Ένωση έχει ε, στενές επαφές με διάφορα υπουργεία αμήνης, εσωτερικών, ε, εξωτερικών, οικονομικών δικαιοσύνης και με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές, την Επιτροπή Προϋπολογισμού, την Επιτροπή Εσωτερικών ε, και ε, βουλευτές ε, του, της Εθνικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης συναντώνται τακτικά και στο παρελθόν είχαμε και πρωτοβουλίες της Ένωσης οι οποίες εκτιμήθηκαν δεόντως από την κυβέρνηση και από το Κοινοβούλιο. Τώρα, σε σχέση με τις μετακινήσεις και τις επαφές με τα ΜΜΕ, κανείς δεν θα ήθελε να πάει ο εκπρόσωπο τη Ένωση και να πει στα ΜΜΕ τα αντίθετα από αυτά που είπε την προηγούμενη μέρα ο υπουργό Αμήνη. Σα δίνω ένα συγκεκριμένο ε, παράδειγμα. Τα ΜΜΕ όμως, τα γερμανικά, θέλουν συνήθως κάποιον ε, που εκπροσωπεί τις ένοπλες δυνάμεις για να προσφέρει την τεχνογνωσία, να παρουσιάζει με ακρίβεια τα προγράμματα και τις αποφάσεις ε, του Υπουργού. Μπορούν λοιπόν εκπρόσωποι και των δύο να δάσκουν σε πολιτικές ε, και μη συζητήσεις σχετικά με το ε, την σταδιοδρομία παραδείγματο χάρη των, ε, του στρατιωτικού προσωπικού ε, ή ακόμη και για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Μετά από μια απόφαση του Γερμανικού Διοικητικού Δικαστηρίου μπορούν επίσης τα μέλη της οργάνωσης να ασχολούνται με θέματα της Ένωσης ενώ φέρουν τη στολή τους. Ε, Γερμανοί στρατιώτες επίσης δικαιούνται να διαδηλώνουν. Έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το 2001, 25.000 εμέλη από τη δική μου οργάνωση και από την ε, αστυνομική συνδικαλιστική οργάνωση διαδήλωσαν ε, στο Βερολίνο κατά ενός νομοσχεδίου σχετικά με μεταρρύθμιση του αξιοδοτικού συστήματος. Ένστολοι διαδήλωσαν και πάλι εδώ πέρα. Ε, οι διαδηλώσεις ενστόλων δεν επιτρέπονται για γενικά πολιτικά ζητήματα που δεν σχετίζονται με τη σταδιοδρομία του στρατιωτικού προσωπικού μόνο όσοι έχουν ένα επαγγελματικό ενδιαφέρον επειδή υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις μπορούν να μετάσχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις ε, και σημειώστε ότι οι Γερμανοί στρατιώτες δεν δικαιούνται να απεργήσουν ούτε και θέλουν ε, να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα διότι γνωρίζουν ότι οφείλουν να υπηρετούν την πατρίδα τους ε, δεν χωρίς αντιλογή ακολουθούν τις διαταγές παραδείγματος χάρη της διοίκησης μπορούν να συζητήσουν ε, τις συνθήκες, ε, την υπηρεσιακή τους κατάσταση με τον Υπουργό, με τον Υφυπουργό, αλλά δεν ε, προβλέπεται απεργία. Επίση, οι Γερμανοί στρατιώτε έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υπηρεσιακή του κατάσταση της μονάδες τους σε επίπεδο Υπουργείου Αμήνη. Τα, αυτά τα δικαιώματα εκτελούνται από δύο ερετά μέλη, δύο πολύ ε, σημαντικών σωμάτων. Πρόκειται για το βασικό Συμβούλιο Προσωπικού και υπάρχει μια τεράστια λέξη τώρα στα γερμανικά που είναι ο τίτλος της δεύτερης ε, ε, του δεύτερου αυτού σημαντικού σώματος ε, είναι μια βασική επιτροπή ουσιαστικά διαπιστευμένων ε, προσώπων, αν θέλετε πρόκειται για ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Αμήνης. Οι υποψήφοι παίρνουν το χρήσμα από τις ενώσεις και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για να εκλεγούν σε αυτά τα δύο τόσο σημαντικά σώματα. Ιδού ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος ε, Αμυράλια που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης ε, Αλληλεγγύης ε, Δικαίου και Προόδου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτές, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, μέλη της Euromil, Από ιταλικής πλευράς προσπαθούμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε μέσω της κοινοτικής νομοθεσίας να διευθετήσουμε το ζήτημα του «Συνεταιρίζεστε» για τους στρατιωτικούς. Έχουμε δει όμως ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλές πολιτικές ευθύνες, οι οποίες μέχρι στιγμής αντιτάσσονται στο αίτημά μας αυτό, στο δικαίωμα του «Συνεταιρίζεστε». Το δικαίωμα του «Συνεταιρίζεστε» έχει ως στόχο να προστατεύσει αστικά τα κοινωνικά δικαιώματα των Ιταλών στρατιωτικών. Και το έτοιμά μας αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από το 1978 όπου είχαμε τον, την νομοθεσία 382 κάθος 78 και συγκεκριμένα το άρθρο 8 το οποίο διευθετεί αυτό το ζήτημα. Στην ουσία αυτό που λέγεται είναι ότι το στρατιωτικό προσωπικό της Ιταλίας δεν μπορεί να δημιουργήσει συνδικαλιστικές οργανώσεις, ούτε μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης, Θεωρείται ότι η δημιουργία οποιοδήποτε σωματείου ή συλλόγου θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να έχει την πρώτερη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Άμυνα. Προκειμένου να κατανοήσουμε τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα, τα οποία προστατεύονται από το Ιταλικό Σύνταγμα, στα άρθρα 18 και 39 συγκεκριμένα, Το 1978 λοιπόν είχαμε τον νόμο 382 κάθετος 78, μετά από έντονες συζητήσεις στην εποχή εκείνη, καταλήξαμε στην νομοθεσία αυτή, όπου συμμετείχαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της εποχής. Βέβαια, στη συζήτηση αυτή είδαμε και το όλο συντηρητικό πνεύμα της εποχής εκείνης, Η μεταρρύθμιση πάντως είναι σαφώς σημαντική, ακριβώς επειδή το εφιστάμενο σύστημα στην Ιταλία αντιτίθεται στα δικαιώματα όπως αυτά προστατεύονται από το Σύνταγμα. Όσον αφορά το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και το Ιταλικό στρατιωτικό προσωπικό, έχουμε την νομοθεσία αυτή λοιπόν του 1978, η οποία αναφέρεται σε κάποια σώματα εκπροσώπησης στα πλαίσια του Ιταλικού στρατού. και αναφέρομαι εδώ πέρα στις ε, εδαφικές στρατιωτικές αρχές της χώρας. Υπάρχει ένα όργανο το οποίο έχει να κάνει με την ε, διαχείριση της δυνατότητας εκπροσώπησης των ε, στρατικών δυνάμεων της Ιταλίας έπρεπε να προβλεφθεί όμω και μια χρηματοδότηση προκειμένου να υπάρχει εκπροσώπηση αυτή και τελικά πολύ γρήγορα συνειδητοποίησαμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μια αυτόνομη εκπροσώπηση των Ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν κάποια εγγενή προβλήματα, κάποιε εγγενεί δυσκολίε στην θέσπιση ε, του σώματος αυτού που θα μπορούσε να εκπροσωπεί τον Ιταλικό στρατό. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 άρχισε να ανανεώνεται το αίτημα αυτό για μεταρρύθμιση, για προάσπιση του δικαιώματος να εταιρίζεστε στα πλαίσια του Ιταλικού στρατού. Προσπαθώντας λοιπόν να ανταποκριθούμε σε ένα γενικότερο συνέστημα για μια νέα νομοθέτηση για τα δικαιώματα αυτά, είδαμε ότι θα έπρεπε να αλλάξει όλο το πολιτικό τοπίο το οποίο ίσχυε τα τελευταία 20 χρόνια. Και όπως σας είπα υπήρχαν, υπήρξαν νέες, νέα αιτήματα μεταρρύθμισης χωρίς όμως αυτά να έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένε πράξεις. Δεν αναφέρομαι εδώ πέρα σε οπορτουνιστικές τάσεις. Πολύ συγκεκριμένα το 1999 είχαμε απόφαση του Σταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας όσον αφορά τη σταγματικότητα της ε, εκπροσώπησης του στρατιωτικού προσωπικού. Πρόκειται λοιπόν για μια απόφαση του Σταγματικού Δικαστηρίου που ελήφθη το 1999. Απόφαση όμως προσπαθούσε να επιλύσει κάποια εσωτερικά προβλήματα του Ιταλικού στρατού. Και πάλι φάνηκε ότι υπήρχαν κάποια γενή προβλήματα στον Ιταλικό στρατό που δεν επέτρεπαν την ε, προάσπιση του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε. Ε, ήδη από την εποχή εκείνη είχαμε πει ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να εφαρμοστούν οι διατάξεις ε, τη του διεθνούς, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση υπαριθμών 449 99 του Σταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, στην οποία τώρα εμείς βασιζόμαστε και βάσει της οποίας απευθυνθήκαμε και στην Euromill. Υπάρχει μάλιστα και ένα κεφάλαιο σε ένα έγγραφο της Euromill το οποίο αναφέρεται σε διάφορες τάσεις αποσιώπησης τέτοιων ετοιμάτων για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι στα πλαίσια του τελικού στρατού. Προσβλέπουμε τώρα σε μια πιο προηγμένη νομοθεσία την οποία προωθεί η Διεθνή Οργάνωση Εργασία και θέλουμε να δούμε αν το πρόβλημά μα μπορεί να επιληθεί σε ένα ευρωπαϊκό, σε ένα κοινοτικό πλαίσιο, στα πλαίσια τη κοινοτική νομοθεσία. και θέλουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις τις οποίες ε, έχουμε μπροστά μας. στο γεγονός ότι ε, ο Ιταλικός στρατός, το Ιταλικό στρατιωτικό προσωπικό δεν έχει καταφέρει να έχει πρόσφαση στο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να υφίστε το δικαίωμα αυτό, ιδίως σε περίοδο ειρήνης. Βασικό μας μέλημα είναι να αποφύγουμε οποιαδήποτε δυσανορμία μπορεί να υπάρχει όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του στρατιωτικού προσωπικού. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη συνεκτικότητα και συνοχή στα πλαίσια της Ιταλικής κοινωνίας. Τα όσα ισχύουν για τους απλούς πολίτες θα πρέπει να ισχύουν και για το στρατιωτικό προσωπικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει η ίδια δομική ομοιογένεια σε όλα τα σώματα εκπροσώπησης προς όφελος και των συμφερόντων του στρατιωτικού προσωπικού. Δεδομένης λοιπόν αυτής της ισορροπίας που πρέπει να επιτύχουμε, προσπαθούμε να εμπνευστούμε από την υπερεθνική διεθνή νομοθεσία, η οποία θα παρήχε τις απαραίτητες εγγύσεις για τα δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν προς τον στρατιωτικό προσωπικό. Αν δείτε πιο συγκεκριμένα, στην σύμβαση του διεθνούς, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπαριθμών 151 78, στη σύμβαση αυτή γίνεται λόγος για την παροχή των απαραίτητων προϋποθέσεων βάσει των οποίων το στρατικό προσωπικό μπορεί να τύχει εκπροσώπησης. Επομένως έχουμε μια σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία εμπνέεται από τα όσα ισχύουν για τους ε, απλούς πολίτες και τα οποία θα μπορούσαν να ισχύουν και για το Ιταλικό στρατικό προσωπικό. Υπάρχει και ένας ε, νόμος της Ιταλικής Δημοκρατίας, υπαριθμών 862 84, που θα μπορούσε να δίνει στο στρατικό προσωπικό τέτοια δικαιώματα με αυτά τα οποία εκχωρεί στο αστυνομικό προσωπικό. Ουσιαστικά η νομοθεσία αυτή, 862 κάθετος 84, μεταφέρει κάποια μέτρα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην Ιταλική νομοθεσία. Αν δούμε όμως ε, τι κάνουν οι νομοθέτες, πως έχουν προσπαθήσει με κάθε τρόπο να παρακάμψουν τα όσα λέγονται στη Σύμβαση 151 78 του ILO. Όπως σας είπα υπάρχουν πάρα πολλοί νομοθέτες οι οποίοι προσπάθησαν να αποφύγουν την μεταφορά στην Ιταλική νομοθεσία της σύμβασης του ILO. Οι επαγγελματικές εγγύσεις που δίνονται από τη Σύμβαση 151 78 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Υποτίθεται ότι ε, ήδη ισχύουν, σύμφωνα τουλάχιστον με εκπροσώπου του Ιταλικού στρατού, υποτίθεται ότι ήδη ισχύουν στα πλαίσια τη ε, Ιταλική νομοθεσία. Χρησιμοποιείται λοιπόν το επιχείρημα αυτό από του νομοθέτε αυτού που αντιτίθενται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε για του στρατιωτικού, και χρησιμοποιούν το επιχείρημα αυτό για να πούν δεν υπάρχει κανένα λόγο να επικαιροποιηθεί η Ιταλική νομοθεσία. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Στερείται όμω βάση στο επιχείρημα αυτό. Είναι διάτριτο. Αρκεί κανεί να δει τη σύμβαση 151-78 τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία, όπου λέγεται ότι ε, οι οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να είναι απόλυτα αυτόνομες και ανεξάρτητες, να μην έχουν καμία σχέση δηλαδή με τις δημόσιες αρχές. Άρθρο 5, παράγραφος 1. Επίσης λέγεται ότι θα πρέπει η οργάνωσή τους να είναι αυτούσια, αυτόνομη. Επίσης γίνεται λόγος για την ε, προστασία των οργανώσεων αυτών από οποιαδήποτε εμπλοκή που θα μπορούσαν να έχουν οι δημόσιες αρχές. Άρθρο 5, παράγραφος 2. Επίσης, γίνεται λόγο στην δυνατότητα επέμβασης από τις δημόσιες αρχές και ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό αν τελικά οι δημόσιες αρχές είναι αυτές οι οποίες δημιουργήσουν σώματα εκπροσώπησης ή αν δοθούν επιδοτήσεις ή άλλου είδους χρηματοδότηση από τις ε, δημόσιες αρχές προς αυτά τα σώματα εκπροσώπησης. Όλα αυτά λέγονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3. Νομίζω ότι όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η ιστορία των λεγόμενων ε, κίτρινων συνδικαλιστικών οργανώσεων που υφίστανται ήδη από την εποχή των απολυταρχικών καθεστώτων ή εξακολουθούν και υφίστανται. Και υπάρχει μία, μπορούμε να πούμε, νοσταλγία ακόμα για αυτές τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από διάφορο στελέχη του Ιταλικού στρατού. Σας εξήγησα λοιπόν ότι από το 1978 έχουν ε, ακουστεί τα πρώτα αιτήματα για αυτό το δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι του Ιταλικού προσωπικού. Έχουμε στη συνέχεια τη σύμβαση του, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και ουσιαστικά η σύμβαση αυτή συνοψίζει τα αιτήματά μας. Αν δούμε τώρα τον στρατικό κανονισμό ο οποίος υφίσταται, σαφώς αυτός δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση τον πλουραλισμό, δεν αφήνει καμία επιλογή προς τους εργαζόμενους, προς τους στρατιωτικούς, ως προς το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και του συνέχεστε. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συνοθήλευμα κανονισμών, το οποίο έχει απλώς επιβληθεί, δεν προβλέπει κανένα περιθώριο ευελιξίας. Το κράτος θεωρείται ότι είναι ο εργοδότης και ουσιαστικά αυτό αποκλείει κάθε έννοια ανεξαρτησίας. Ουσιαστικά δεν δίνεται κανένα δικαίωμα συνεταιρίζεστε, καμία ελευθερία προς το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και του συνέχερστε. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια ανεξαρτησία από τις δημόσιες αρχές. Αρκεί να δει κανεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του κυρίου Μπερδουσκόνη ε, πενεύει σε διάφορα στρατιωτικά ζητήματα. και είδαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί στρατιωτικοί οι οποίοι μετακινήθηκαν από τη θέση τους από τη μία μέρα στην άλλη και δεν υπήρξε καμία αντίδραση σε εθνικό επίπεδο. Καμία αντιτιθέμενη φωνή δεν ακούστηκε. Η παρέμβαση λοιπόν της κυβέρνησης του κράτους αντιτίθεται στις δημοκρατικές αρχές που θα πρέπει φυσιολογικά να διέπουν τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργεί ο Ιταλικός ε, στρατός. Βλέπουμε ότι η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί και ουσιαστικά χέρι της συνένεσης διαφόρων πολιτικών ομάδων και πολιτικών κομμάτων στη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου σωστή καθότι δεν παρέχει καμία ελευθερία στο στρατιωτικό προσωπικό. το οποίο ουσιαστικά παραμένει δεσμευμένο στις δημόσιες αρχές. Σαφώς όμως τα πράγματα εξελίσσονται. Έχουμε πλέον τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε όλο και περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία προασπίζονται τυχαίων προστασίες, με συγχωρείτε, στα πλαίσια τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εμείς προσβλέπουμε όλο και περισσότερο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά στην περίοδο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και θέλουμε να δούμε πώς θα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, να υλοποιηθεί στην πράξη η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι μέσω των μέσων αυτών θα καταφέρουμε ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε τον ιδεολογικό συντηρητισμό που έχουμε στην Ιταλία και που έχει αποτελέσει τροχοπέδι σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει στο παρελθόν. Πιστεύω ότι το ASSODIPRO θα συνεχίσει την εργασία του και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε τουλάχιστον το 2012, το επόμενο έτος, να επιτύχουμε ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Έχουμε ήδη τα πρώτα θετικά δείγματα τα οποία καταδεικνύουν ότι οι καιροί αλλάζουν. Σαφώς υπάρχουν ε, συντεχνιακά ακόμα συμφέροντα τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Πιστεύω πάντως ότι αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα τροποποιηθούν προς το καλύτερο και ενδεχομένως τελικά να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε το συντομότερο δυνατό μία πολιτική προστασία για τα βασικά αυτά δικαιώματα τα οποία προωθούμε. Προσβλέπουμε λοιπόν σε οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε να έχουμε από εσά, Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να ακούσουμε ερωτήσεις ή σχόλια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Πρόεδρε, για μένα είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε με προσοχή αυτή την ακρόαση, ιδιαίτερα επειδή η υποεπιτροπή έχει τώρα την ευκαιρία να συντάξει μία έξεση μαζί με την Euromil Και δεύτερον, επειδή πρόκειται για το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και για να, για να μπορούμε να ενημερωθούμε, να συλλέξουμε πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε το έργο της ε, ολοκλήρωσης και της ε, εφαρμογής αυτού του δικαιώματος σε όλη την Ευρώπη. Ακούσαμε πολλά ε, σχόλια ε, αλλά και σημειώσαμε διάφορες ελλείψεις ακόμα και πολλούς περιορισμούς στα δικαιώματα. Ιδίως στο γεωγραφικό χάρτη βλέπουμε μεγάλες ανισότητες. Αυτό μας ε, πρέπει να μας δώσει ε, τη δυνατότητα και το έναυσμα να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο ως ευρωβουλευτές. Αυτή τη στιγμή βέβαια αντιμετωπίζουμε μια καινούργια πραγματικότητα ε, και σε πολιτικό επίπεδο αλλά έχουμε και μεγάλες προκλήσεις στο νομικό πλαίσιο που αντιμετωπίζουμε και στις αρμοδιότητες δεν υπάρχει ένα ενοποιημένο καθεστώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ορισμό αυτού του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε. Δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα αυτή και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Πολλές φορές μελετήσαμε το πρόβλημα αυτό και η Κομισιόν πάντοτε μας δίνει την ίδια απάντηση. Είναι εκτός αρμοδιοτήτων μας. Όμως, ε, το νομικό πλαίσιο έχει εξελιχθεί. Εδώ πρόκειται και για το χάρτη των, ανθρωπίνων, των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, πρέπει να γίνουν σεβαστές αυτές οι διατάξεις και πρέπει να δούμε εάν δεν έχει μεγαλώσει, δεν έχει δυναμώσει η ισχύς αυτού του χάρτη και αυτών των δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά εδώ βασικά μας ενδιαφέρει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουμε αυτόν τον χάρτη ο οποίος δεν οδηγεί αυτόματα σε αρμοδιότητες ε, νομικής φύσεως. Και κανένας δεν το ισχυρίζεται αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως ε, πρέπει να εργαστούμε για μια πιο συνεπή και συνεκτική εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και να συντονίσουμε ε, τα δικαιώματα αυτά και τις διατάξεις αυτές ε, ως βάση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Και αυτά τα βασικά δικαιώματα συμπεριλαμβάνουν και το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Αυτό ισχύει σε όλες τις οργανώσεις ή τους οργανισμούς εργασίας. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτές οι δύο διαφορετικές νομικές βάσεις, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε κατά πόσο τα εθνικά νομικά πλαίσια προσφέρουν ή εξασφαλίζουν αυτό το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε ή δεν το εξασφαλίζουν. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση ε, σε κάθε χώρα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για την Ιταλική εσωτερική κατάσταση, όμως πρέπει να πω ότι οι στρατιώτες δεν μπορούν από μόνοι τους να τα εξασφαλίσουν όλα αυτά, όμως σιγά σιγά έχουν σημειωθεί εξελίξεις που βοηθούν την ελεύθερη έκφραση των μελών των ενόπλων δυνάμεων. Στην Ιταλία βεβαίως μόνο με τη ρητή άδεια των προϊσταμένων. Και αυτό είναι κατά του, ανθρωπ, των, του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, δεν λέω, αλλά ε, έχουν, ε, έχουν γίνει και ποινικέ διώξεις εναντίον μελών των ενόπλων δυνάμεων επειδή ακριβώς φύρμωσαν αυτό το δικαίωμα ή συγκεντρώθηκαν κάπου ε, δεν, μιλάω βέβαια για παράνομες ε, ε, συνελεύσεις ή, ή παράνομες ενώσεις με σκοπό να βλάψουν την εθνική ασφάλεια της Ιταλίας. Αλλά για την Ιταλία είναι πολύ, σημαντικό, πολύ σημαντική η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ε, σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το ζήτημα. Και ας μην ξεχνάμε ότι εδώ μέσα στο σώμα αυτό αναπτύσσονται οι βέλτιστες πρακτικές και πάνω σε αυτές πρέπει να βασιστούμε. Καταρχάς λοιπόν μπορούμε με ψηφίσματα ή με προφορικές ερωτήσεις ή με άλλα κείμετα, κείμενα να συνεργαστούμε με άλλους συναδέλφους, παραδείγματο χάρη με τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και να ζητήσουμε επίμονα την εφαρμογή αυτών των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Από την άλλη πλευρά πρέπει μέσω νέων, νέων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας ε, οι πράξεων να προσπαθήσουμε και με τα μέσα ή τις πράξεις που διατίθενται από πλευράς Κομισιόν να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα όλες, όλα τα κράτη-μέλη, ιδίω να πιέσουμε τις χώρες εκείνες όπου δεν αναγνωρίζονται. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε ε, την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτών στις ένοπλες δυνάμεις σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ κύριος Γκάιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά ε, θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφός μου, κύριος Γκουαλτιέρη. Όλα αυτά τα οποία είπε θα πρέπει να τα μελετήσουμε. Πιστεύω ότι από αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα είναι σαφής ε, ο στόχος μας. Αφενός θέλουμε, ε, συμφωνούμε δηλαδή στη διαπίστωση ότι ο στρατιώτης είναι ένας ένστολος πολίτης και έχει όλα τα δικαιώματα και από την άλλη πλευρά ε, πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδυναμώνεται ούτε διακυβεύεται η τάξη και η ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων, η ιεραρχία, η πεισαρχία κλπ. με τη συγκρότηση τέτοιων ε, ενώσεων ή συνδέσμων. Επίσης, ένας υπουργός άμυνας ή ένας αρχηγός επιτελείου ε, μπορεί να τον βολεύει ιδιαίτερα να μην υπάρχει μία ε, τέτοια οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων ε, έτσι ώστε να μην γίνει καμία φασαρία ας πούμε είναι άλλο πράγμα να παραπονιέται ένα στρατιώτη ότι η στολή του δεν είναι σωστή και στα μέτρα του και άλλο να γίνονται να ακούγονται κατηγορίες ότι λόγω των ελληπών στολών ή των, του κακού εξοπλισμού διακυβεύεται η ζωή και η ασφάλεια των ε, στρατιωτών και έτσι ας πούμε οδηγούνται σε ατυχήματα και δίσανα τη φόρα. Άλλο τον άλλο τ' άλλο. Αλλά εδώ οι συνεταιριζόμενοι, οι συνδικαλιστές δεν θέλουν να υπονομεύσουν τις ένοπλες δυνάμεις, απλώς θέλουν να βελτιώσουν ε, τη θέση τους και την κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις έτσι ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά ε, τον ε, σκοπό τους και να εκτελέσουν καλύτερα το καθήκον τους θα ε, μπορούμε, ας πούμε, θα, μπορούν να συζητήσουν ε, την βελτίωση ε, των συνθήκων εργασίας, η υπηρεσίας, των, ε, της άδειας, της παρεχόμενης άδειας, της, του συνδυασμού της στρατιωτικής επαγγελματικής ζωής με την οικογενειακή ζωή και πολλά άλλα θέματα. Γι' αυτό ίσως ε, υπάρχουν ε, ορισμένες καλύτερες ελπίδες ε, τώρα, οι προσδοκίες για τους Ιταλούς φίλους μας με την αλλαγή της κυβέρνησης. Είναι βέβαια δύσκολο να παραιτηθεί κανείς από παλιές συνήθειες και από φοβίες που υπάρχουν, διότι πολλοί ακόμα πιστεύουν ότι κάθε τέτοιο δικαίωμα θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, αναταραχές και φασαρίες. κάποτε είχα και εγώ την εμπειρία ε, την πρώτη εβδομάδα που υπηρέτησα στον γερμανικό στρατό μου έδωσαν αμέσω μία αίτηση να συμπληρώσω για να συμμετάσχω στην κατάλληλη ας πούμε ένωση των, ε, που μπορούσα να υπαχθώ εγώ και μέσω της ενώσεως αυτής είχα και εγώ το δικαίωμα να, παρα, να παραπονεθώ ή να γύρω διάφορα αιτήματα. Εγώ από τότε παρέμεινα και μέλος του Συνδέσμου Ενόπλων Δυνάμεων της Γερμανίας, του στρατιωτικού συνδέσμου, από, για λόγους αρχής αλλά είναι πάρα πολύ σωστό νομίζω να υπάρχει πάντοτε ένας φορέας με τον οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει τα προβλήματα που προκύπτουν. Ε, εγώ είχα αυτή την εμπειρία που σας είπα κατά την περίοδο της θητείας μου και πιστεύω ότι αυτό το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και οι συναφείς ε, ενώσεις μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στη διευθέτηση προβλημάτων. Αντί να γύρει ο κάθε ε, στρατιώτης, ας πούμε, ε, μέσω ενός αιτήματο, ε, να παρακαλεί δηλαδή για, για την επίλυση ενός προβλήματος. Πιστεύω λοιπόν ότι και ε, οι Ιταλοί φίλοι μας θα μπορέσουν να επιφοληθούν στο μέλλον και για αυτό το στόχο εξυπηρετεί και η σημερινή μας ακρόαση. Από τη μία πλευρά στο ευρωπαϊκό επίπεδο να υποστηρίξουμε και να δηλώσουμε την υποστήριξή μας στους συναδέλφους της ε, Euromil ότι υποστηρίζουμε και ηθικά και πολιτικά αυτές ε, τις ενώσεις και αυτή τη διαδικασία και δεύτερον να ξεκινήσουμε μία αντικειμενική συζήτηση, ένα διάλογο και ενδεχομένως να βρούμε νέες λύσεις, νέες προσεγγίσεις με τη συζήτηση με τον νέο Υπουργό Αμήνης ή με τους νέους αρμόδιους ε, φορείς. Πιστεύω ότι προσφέρεται αυτή η ευκαιρία τώρα μιας ε, κοινή συζήτηση ε, διότι μέσω μιας ε, τέτοιας ένωσης, ενός τέτοιου φορέα, μπορεί να συζητήσουμε πάρα πολλά στρατιωτικά θέματα ο Υπουργός, ε, παραδείγματο χάρη, μέσω των ε, φορέων αυτών, των στρατιωτικών ε, ενώσεων, μπορεί να υποβάλει και προτάσεις στον Υπουργό Οικονομικών. Τα διάφορα αιτήματα δηλαδή μπορεί να περνάνε από τις ενώσεις, τους συνδέσμους αυτούς στον Υπουργό Άμυνας και συνεχεία στους άλλους συναρμόδιους υπουργούς. Είναι ένα κανάλι επικοινωνίας σημαντικό και χωρίς να είναι κανείς εγκυλωμένος στις παραδοσιακές δομές και φοβίες μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως τους Ιταλούς συναδέλφους και να τους ε, στηρίξουμε είτε πολιτικά είτε μέσω των νομίμων διοικητικών δομών, μέσω των νομίμων οργανώσεων, να τους προσφέρουμε κάθε υποστήριξη στα ε, αιτήματά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, κυρίους για τις, παρουσιάσει για τις παρουσιάσεις που κάνανε δώσαν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία ε, για την κατάσταση σε συγκεκριμένες χώρες. Εν τούτης, θα ήθελα να ε, σημειώσω κάποιες σκέψεις που σίγουρα δεν ε, θα βρούνε την σύμφωνη γνώμη αλλά χρειάζεται για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ και εγώ με το γεγονός ότι η ένστολη θα έπρεπε να είναι πολίτες με τα ίδια δικαιώματα όπως έχουν και άλλοι πολίτες. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, ποτέ δεν έγινε και όσες ενώσεις ε, και να κάνουμε στις ένοπλες δυνάμεις ποτέ δεν θα συμβεί. Είναι άγραφος νόμος, αλλά είναι αλήθεια αυτό, ότι σε όλους τους καπιταλιστικούς στρατούς δεν μπορεί να έχουν πολιτική γνώμη. Δεν θα βρείτε κανένα στρατό που να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα οι εφημερίδες εφημερίδες ενός κομμουνιστικού κόμματος ή ξέρω εγώ μια αριστερή εφημερίδα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ω εκ τούτου καλό είναι ορισμένα πράγματα να είναι ε, σε συγκεκριμένα πλαίσια. Το δεύτερο που ήθελα να σημειώσω και να εκφράσω την ανησυχία μου για το γεγονός ότι γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια τάση όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα ενάντια στις συλλογικές μορφές οργάνωσης και διαπραγμάτευσης. Ας πούμε στην Ελλάδα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Για ποιες συλλογικές διαδικασίες θα μπορούσε κανείς να μιλήσει γενικότερα. Ε, επίσης, νομίζω ότι δεν ε, αναλύεται σωστά ο ρόλος και οι τεράστιες ευθύνες, αλλά όχι και τα δικαιώματα που ζητιέται σήμερα, ζητιούνται σήμερα από τους ένστολους από τα αστικά κράτη και εξηγούμε. Η κατάσταση η οποία περιγράφθηκε παραδείγματο χάρη για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των ενστόλων στη Γερμανία ε, ανταποκρινόταν σε μια εποχή όπου ο γερμανικός στρατός ήταν περιορισμένος αυστηρά σε ρόλο υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας του και δεν είχε κανένα ρόλο όσον αφορά το εσωτερικό της χώρας, την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Ξέρουμε όμως ότι μετά τη δεκαετία του 90 όλοι οι στρατοί, όχι μόνο ο γερμανικός στρατός, και ο ελληνικός και ο ιταλικός και ο ισπανικός, όλοι οι στρατοί, έχουν ε, αλλάξει το ρόλο τους και έχουν γίνει κυρίως στρατοί με δράση στο εξωτερικό, σε εμπεριαλιστικούς πολέμους, είτε είναι στο Κόσοβο, είτε είναι στο Αφγανιστάν, είτε είναι στο Πακιστάν ή αλλού. Είναι δυνατόν οι ενώσει των στρατιωτικών να μην έχουν άποψη και το ίδιο συμβαίνει και για το εσωτερικό των χωρών βεβαίως. Ξέρετε δεν υπάρχει καμία μεγάλη διεθνή συνάντηση όπου να μην επιστρατεύεται και ο στρατός. Ξέρετε επίσης ότι υπάρχουν νόμοι που επιτρέπουν την δράση του στρατού και για την πάταξη ε, πώς το εσωτερικής ε, αναταραχής. Στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη έχει γίνει άσκηση πρόσφατα ε, των Euro Battle Groups για ε, καταστολή διαδήλωσης αντιπολεμικής. Συνεπώς το λέω. Οι ενώσει των στρατιωτικών δεν μπορεί να μείνουν εκ των πραγμάτων, αν θέλουμε να λέμε αυτό που λέμε, ότι οι ένστολοι είναι και πολίτες ένστολοι, δεν μπορεί να μείνουν μόνο με συνδικαλιστικές λειτουργίες και συνδικαλιστικές δράσεις. Παραδείγματος χάρη κύριε Πρόεδρε, αυτές τις μέρες προχθές έγινε αυτό το, το, το, το, το απαράδεκτο και αυτή η δολοφονική πράξη του ΝΑΤΟ στο Πακιστάν. Έτσι δεν είναι, όλοι την ξέρουμε. Παράν. Αν εγώ δεν είδα κανένα, καμία ένωση ενστόλων που να διαμαρτύρεται για αυτό το πράγμα. Ούτε τώρα ούτε στο παρελθόν. Είναι δυνατόν να συνεχίσετε αυτή η κατάσταση. Ε, Προφανέ ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Γι' αυτό το λέω κιόλα ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έγινε. Ε, εγώ υποστηρίζω και τάσουμε αναφαντών υπέρ της ανάγκης ε, της οργάνωσης των, ε, των ε, στρατιωτών γιατί πράγματι έχουν δικαιώματα όμως πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για τα πολιτικά τους δικαιώματα. Δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή να, να, να τους... γιατί ξέρουμε ότι όλοι έχουν και σκέψεις και απόψεις και, και δυνατότητες. Παραδείγματο χάρη θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που υπόθηκε ότι ο συνδικαλισμό στο στρατό δεν είναι εμπόδιο ούτε για την πειθαρχία ούτε για την, επιχειρηματικότητα, για την επιχειρησιακή του δράση. Εξάλλου να θυμίσω, τα Wikileaks δεν προήλθαν επειδή στον Αμερικάνικο στρατό υπήρχε συνδικαλισμός. Έτσι δεν είναι. Δεν υπήρχε τίποτα. Και παρόλα αυτά βγήκαν τόσα πράγματα ε, στη φόρα. Επίσης δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει σε ένοπλε δυνάμει των ευρωπαϊκών χωρών τη στιγμή που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να αφαιρεθούμε από αυτό το πράγμα. Είναι άραγε τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι στρατοί είναι και μέλη του ΝΑΤΟ και ε, αυτό έχει οπωσδήποτε σχέση και με, αυτή την, ε, και με αυτό το ε, ζήτημα. Κλείνοντα, έχει τεράστια σημασία η διαπαιδαγωγή στι ενόπλε δυνάμει. Και από τη στιγμή που οι ένοπλε δυνάμει σήμερα διαπαιδαγωγούνται και για επιχειρήσει εκ των συνόρων, επιθετικέ και εντό συνόρων, μη σα κάνει εντύπωση να έχουμε τέτοιου είδου επεισόδια που δυστυχώ έχουν συμβεί, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πριν μια εβδομάδα στην Ελλάδα, όπου μέσα στο ελληνικό στράτευμα, είναι βέβαια μια, ε, μια μεμονωμένη περίπτωση, ε, έγινε προσπάθεια από ε, ε εκπαιδευμένους αξιωματικούς να επαναφέρουν με έναν τρόπο τη στρατιωτική χούντα, τη, τη δικτατορία. Αυτό για μας έχει σχέση με, με το γενικότερο κλίμα που υπάρχει και γι' αυτό το λόγο κλείνω λέγοντας ότι θα έπρεπε οι ένστολοι να έχουν και πολιτικά δικαιώματα και οι οργανώσεις τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Ε, θα ακολουθήσουμε την ίδια σύρα. Ε, σειρά. Ο κύριος Τζέικοφ θα πάρει πρώτος το λόγο για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις ε, παρατηρήσεις που ακούσαμε. Θα ήθελα εν συντομία να σχολιάσω όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρήσουμε το εξή. Όταν οργανώνονται οι στρατιωτικοί ενώσει ή συνδικαλιστικέ οργανώσει, ε, τότε δέχονται χωρί κανένα πρόβλημα το ότι υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα δικαιώματά τους καμία, καμία στρατιωτική συνδικαλιστική οργάνωση ή ένωση δεν το προβλέπει αυτό. Ίσως κάποιοι μεμονωμένοι στρατιώτες, τέλος πάντων σωματεία, ενώσεις και οργανώσεις δεν το προβλέπουν αυτό. Δεν, δεν ζητούν καν το δικαίωμα ε, του Απέργεν και στην Ευρώπη. Έχουμε κάποιες χώρες όπου προβλέπεται το δικαίωμα της απεργίας, ακόμη και για τους στρατιωτικούς, ποτέ όμως δεν έχει γίνει χρήση αυτού του δικαιώματος. Πέρα από μια διαδήλωση δεν έχει σημειωθεί ποτέ απεργία από στρατιωτικούς. Οι στρατιωτικές ενώσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζουν μια χαρά και δέχονται το ότι ε, σε επιχειρησιακό επίπεδο οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί άμυνας, ε, πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις ή το Γενικό Επιτελείο. Τώρα, σε σχέση με την εκτέλεση ορισμένων επιχειρήσεων και την ίδια την επιχείρηση, μπορούν να κάνουν κάποια σχόλια. Δίνω ένα παράδειγμα. Υπάρχει η απόφαση να μεταβούν, δεν ξέρω εγώ πού, οι στρατιώτες, απόφαση που λήφθη από μια κυβέρνηση, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα σχόλιο θα εκτελεστεί αυτή η διαταγή. Εμείς όταν ισχυριζόμαστε ότι οι στρατιώτε αποφαση που ληφθη απο μια κυβερνηση χωρις κανενα προβλημα χωρις κανενα σχολιο θα εκτελεστει αυτη η διαταγη Εμεί, οταν ισχυριζομαστε τουλάχιστον να έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται, δηλαδή συγγνώμη, να ενημερώνουν τη στρατιωτική ηγεσία, να ενημερώνουν <clears throat> την ε, πολιτική ηγεσία για τα ε, προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν. Ε, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ευημερία των στρατιωτών. Λοιπόν, οι στρατιωτικοί μπορούν να ενημερώσουν την πολιτική ηγεσία. Ο κύριος Γκάλερ νομίζω μας είπε ότι δεν προβλέπονται ενώσει, ε, δεν προβλέπονται συνδικαλιστικές οργανώσεις σε βάση του Υπουργού Άμυνα Μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά ε, από τη δική μου εμπειρία ξέρω πως ε, οι ενώσεις δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεμονωμένων στρατιωτών και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δική μας οργάνωση ή η συνδικαλιστική οργάνωση που υπάρχει στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία ή στην Ιρλανδία συχνά ε, συνεργάζονται με την, στρατιωτική, με την πολιτική ηγεσία, με την κυβέρνηση για το καλό ε, των ε, ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχουν στιγμές όπου θα γίνουν καταγγελίες από πλευράς των στρατιωτών. Θα προκύψει διάσταση απόψεων, αλλά και 27 στρατηγούς να βάλετε μαζί πάλι θα υπάρξει διάσταση απόψεων. Εσωτερικά θα πούνε όλοι ότι εξωτερικά προς τα έξω, προς τον έξω κόσμο θα πούνε όλοι ότι συμφωνούν, αλλά θα διαφωνήσουν ε, εσωτερικά. Και άρα θα προκύψει διάσταση απόψε ανάμεσα στο στρατιωτικό προσωπικό και την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνα, παραδείγματο χάρη. Αλλά ξαναλέω, εξυπηρετούμε το γενικό καλό, όχι μόνο το καλό των στρατιωτών, το καλό των ενόπλων δυνάμεων. Ε, Σχεδόν το δικαίωμα το συνεταιρίζεστε. Ε, δεν είναι το μόνο, μπορούμε να συζητήσουμε και για άλλα δικαιώματα, ε, για δικαίωμα για δίκη, δίκη, δικαίωμα έκφρασης, δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα οργανώσεων τύπου, μάλλον θεσμών τύπου διαμεσολαβητή κτλ. Αλλά δεν εμπίπτουν αυτά στην σημερινή μας συνεδρίαση. το, αυτό το πιο ωφέλιμο που έχουμε να κάνουμε να ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση. Έχει ξεκινήσει επίσης ε, διάλογος ε, για ολοκλήρωση για ενοποίηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, για συγχρονισμό της δράσης τους σε κάποιες χώρες. Το μόνο θετικό της ε, οικονομικής κρίσης είναι ότι υποχρεούνται πολύ περισσότερο σχέση με το παρελθόν να συνεργαστούν οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις. Όμως, πώς θα το εξηγήσουμε στον κόσμο, δηλαδή ότι αν αρχίσουν να συνεργάζονται ένα και περισσότερο ε, οι ένοπλες δυνάμεις, όταν πάμε στο Ιγκαμπούλ, στο αεροδρόμιο, 35 έθνη εργάζονται στο ίδιο ε, αεροδρόμιο. Πώς να εξηγήσετε όλοι, ότι όλοι έχουν ουσιαστικά τα ίδια καθήκοντα και προσωπούν ε, τους ίδιους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, αλλά έχουν εντελώς διαφορετικά δικαιώματα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στους στρατιώτες. Και ε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση θα βρει την υποστήριξή μας. Προσπαθούμε να πείσουμε τους υπουργού Άμυνα, ορισμένες φορές τα καταφέρνουμε, προσπαθούμε ε, να πείσουμε τους ε, στρατηγούς, ε, κυρίως να αποστρατεία πείθονται και Ε, αλλά σας, και ε, δέχονται ε, να μας υποστηρίξουν στη δράση μας, αλλά κυρίως τα εναποστρατεία, όπως σας είπα. Ο, τα εθνικά κοινοβούλια είναι αυτά που μας βοηθούν περισσότερο από όλους. Αυτά πρέπει να πείσουμε. Να, μια νίκη που είχαμε είναι στην Ισπανία για την αναγνώριση του δικαιώματο του συνεταιρίζεσαι. Δεν θα ισχυριστώ ότι χάρη σε εμά έγινε αυτό, αλλά πόσε φορέ πήγαμε εκεί να μιλήσουμε ακόμη και τέσσερι φορέ τη μέρα με εκπροσώπους όλων των πολιτικών παρατάξεων, επισκεφτήκαμε κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Τέλος πάντων, εστεύθη μια επιτυχία αυτό το, ε, αυτή η απόπειρά μα και αναγνωρίζεται, κατοχυρώνεται πλέον αυτό το δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι στην Ισπανία. Λοιπόν, η συνεργασία είναι προ όφελο και του στρατιωτικού προσωπικού και των κυβερνήσεων κυβερνήσεων. Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι η Πολωνία που αντέγραψε κάποια αποσπάσματα τη νομοθεσία, ενό νομοσχεδίου μάλλον που ήταν υποσυζήτηση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Πήραν αυτά τα αποσπάσματα, τα πήγανε στην Πολωνία και τα κατέθεσαν στην Πολωνική Βουλή και τελικά ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία. Ένα άλλο ένα παράδειγμα ε, που καταδεικνύει ότι είναι δυνατόν ε, να ε, τα καταφέρουμε να συνεργαστούμε. Ε, για την Ιταλία δυστυχώς ε, χρησιμοποιήθηκε ως αρνητικό παράδειγμα. Σήμερα τώρα θα αρχίσουμε ε, τις συνομιλίες με το έναν άβαρχο που είναι ο νέος Υπουργός Άμυνας. και δεδομένων αυτών των ιδιωτήτων του ε, πρώην Ναύαρχος Νίνη υπουργό Άμυνα, ε, δύσκολα θα δεχτεί τις θέσεις μας αλλά δεν μπορούμε και να προδικάζουμε το πώς θα τοποθετηθεί κάποιο, θα προσπαθήσουμε συχνά. Το πρόγραμμα είναι το εξή ότι όταν ε, ρωτάμε τους Υπουργού Άμυνα ή τους αρχηγούς των επιτελείων γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί και αυτοί να ανήκουν σε δικαλιστικέ οργανώσεις και σε ενώσεις. Μας λένε ότι το πρόβλημα είναι να πείσουν τους υπολείπους στα, ε, στο ΓΕΣΕ ή στη ή στη, τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Άμυνας ε, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για εθνικά ζητήματα, εθνικές αρμοδιότητες, δεν θέλουν να εμπλακούν καν σε μια τέτοια συζήτηση. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους Πορτογάλους συναδελφούς μας, παραδείγματο χάρη, ε, και στην αρχή ήταν άκαρπες οι προσπάθειές μας, μετά από λίγα χρόνια πάντως και, και τα καταφέραμε. Οι στρατιώτες έχουν πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα, πολύ συγκεκριμένη αποστολή και χρειάζεται συζήτηση όλα τα δικαιώματα θεωρητικά μπορούν να εκχωρηθούν στους στρατιώτες, αλλά οι ίδιοι φυσικά δέχονται τους περιορισμούς και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι διάζουσα η περίπτωσή τους και ότι δεν εργάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών στο ταχυδρομείο. Οι περισσότεροι, και το τονίζω, οι περισσότεροι ε, ε, κατατάχθηκαν ε, οικειοθελώς και θέλουν να επιτελέσουν αυτά τα καθήκοντα, αναγνωρίζουν, δέχονται τους περιορισμούς, αλλά αλλά ε, να αναγνωρίζει κανεί του περιορισμού, χρειάζεται διάλογο, χρειάζεται συζήτηση. Αν δεν έχουμε διάλογο, μάλλον για να γίνει διάλογο πρέπει να γνωρίζετε ποιο είναι ο συνομιλωτή σα. Αλλιώ ποτέ δεν πρόκειται να βρείτε μία λύση. Τέλο. Το να μην υπάρχουν τέτοιες ενώσεις ε, ε, έχει τα εξής αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη στην Ιταλία δεν υπάρχει καμία τέτοια ένωση που να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των στρατιωτών, αλλά ας το δείτε και υπό ένα από μια ευρύτερη οπτική γωνία. Δεν είναι το θέμα τη συνεδρίασή μα. Θέλω μόνο εν παρόδο να αναφερθώ σε μια έκθεση κάποιων που εμπιστεύτηκαν τη Σαρδινία για να επισκεφτούν ένα κέντρο ε, αποθήκευσης, απόρριψης πυρομαχικών και ελέγχου ε, οπλικών συστημάτων. Αλλά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Είναι μόνοι τους εγκαταλειμμένοι στρατιώτες εκεί. Να το αποτέλεσμα του να μην υπάρχει καμία τέτοια επαγγελματική ένωση ε, και οι στρατιώτες ε, ή οι οικογένειες των στρατιωτών που στο μεταξύ πέθαναν ε, λόγω όλων αυτών διαμαρτύρονται αλλά κανείς δεν τους ακούει. Και γι' αυτό είναι αγαστό, ή μάλλον είναι επιθυμητό να υπάρχει στενή συνεργασία και διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους αυτών των ενώσεων και την πολιτική ηγεσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα σχολιάσω σύντομα την παρέμβαση του κυρίου Αγκουράκη. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ του να χαίρει κανείς του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε και των ε, ε, ενεργειών που έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Εμείς ε, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και αυτό καλύπτει την, την ελεύθερη έκφραση συνθηκών εργασίας. Καμία σχέση με πολιτικές ε, δηλώσεις. Οι Γερμανοί στρατιώτες επιτρέπεται να είναι μέλη πολιτικών κομμάτων αλλά δεν τους επιτρέπεται να ξεκινήσουν πολιτική συζήτηση στην καθημερινή τους εργασία ε, στα στρατόπεδα που υπηρετούν. Μπορεί στον ελεύθερο χρόνο τους να κάνουν πολιτικές συζητήσεις, αλλά όχι κατά την περίοδο της εργασίας τους. Σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Γκάλας, Βεβαίω, ε, ο Υπουργό Αμήνη, το Γενικό Επιτελείο, η Ένωση Συνδέσμων και οργανισμών, τέτοιων οργανισμών δεν έχουν πάντοτε την ίδια άποψη και την ίδια γνώμη. Ο καθένα έχει το δικό του καταστατικό, τους δικούς του κανόνε εργασίας. Και ε, συνήθως ε, οι σύνδεσμοι αυτοί, οι στατιωτικοί σύνδεσμοι ζητούν πάντοτε περισσότερα από αυτά που ο Άμυνα ε, είναι πρόθυμο να προσφέρει. Όμως όπως είπε ο κύριος Γκάλα, στην πολιτική συζήτηση για το ε, στρατιωτικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό άμυνας, ο, οι αρμόδιοι υπουργοί μπορούν να πάρουν πολλές πληροφορίες από αυτούς τους στρατιωτικούς ε, συνδέσμους. Παραδείγματο χάρη, ανάγκες που υπάρχουν στο θέματα ανάπτυξης δυνάμεων ή ανάγκες που υπάρχουν στον ε, στρατιωτικό εξοπλισμό. Ορισμένες φορές στη Γερμανία ε, βουλευτές σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των στρατιωτικών συνδέσμων κατάφεραν να λύσουν προβλήματα τα οποία ήταν αντίθετα με την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή να λύσουν άλλα ζητήματα με πολύ καλά αποτελέσματα. Βεβαίως ε, πρέπει όλες αυτές οι διαδικασίες και να είναι διαφανείς έτσι ώστε οι Ιταλοί μας συνάδελφοι και το Ιταλικό Κοινοβούλιο να μην φοβούνται ε, τη δημιουργία ή τη σύσταση αυτών των συνδέσμων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ουσιαστικά, συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους μου Α, ένα λεπτό, διακόπτει ο κύριος Γκαουτιέρη. Έχω μία άλλη συγκεκριμένη ερώτηση. Θέλω να διευκρινίσω ότι ε, όσον αφορά τα δικαιώματα στους ιδιωτικούς συνδέσμους και εκεί όπου υπάρχουν διαφορές με το γερμανικό μοντέλο, μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι διαφορές με το γερμανικό μοντέλο. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μιράγκλια. Κοιτάξτε, αυτό το σύστημα ε, στην Ιταλία συνοδεύεται από, ένα, από μια διαδικασία εκλογών ε, και πρέπει να αναλύσουμε αν αυτές οι εκλογικές διαδικασίες για την ε, εκλογή των εκπροσώπων είναι δημοκρατική δεδομένου ότι το εκλογικό σύστημα είναι εξαιρετικά κεντρικοποιημένο και ξέρουμε ότι στην Ιταλία, στις άνοπλες ε, δυνάμεις, οι περισσότεροι στρατιώτες είναι 200.000. 200.000 στρατιώτες και αξιωματικοί. Υπάρχουν όμως και άλλες ενώσεις ε, αξιωματικών ή εθελοντών και αυτή τη στιγμή η στρατιωτική εκπροσώπησή μας έχει συγκερασμένες αρμοδιότητες αλλά δεν είναι στην ισόβαθμη με τους ε, πολίτες. Εδώ έχουμε δύο πτυχές που πρέπει να λύσουμε. Είναι ισόβαθμοι με τις πολιτικές ε, αστικές οργανώσεις, η ε, στρατιωτικοί σύνδεσμοι ή όχι. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων εκπροσωπείται καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Ε, αλλά οι αρχηγοί των επιτελείων φοβούνται την ε, παραχώρηση επιπλέον εξουσιών. Και πρόσφατα έχουμε παραδείγματα τα οποία μας ε, στεναχωρούν ιδιαίτερα ε, διότι βλέπουμε μια σκλήρινση της ε, στάσης ε, στα επιτελεία και φοβούμεθα μήπως πιέσουν τη νέα κυβέρνηση να αλλάξει το νομικό πλαίσιο και τον εκλογικό κανονισμό. Οπότε μπορεί ενδεχομένως να υποστηρίξουν ε, την εκλογή εκπροσώπων οι οποίοι πάνε με τα νερά των ε, προϊσταμένων, με τα νερά των επιτελαρχών και δεν δημιουργούν προβλήματα. Δεν πιέζουν δηλαδή για πρόοδο. Η κυβέρνηση έχει παρέμβει πολλές φορές σε αυτά τα ζητήματα όσον αφορά την ε, οργάνωση εκλογικών διαδικασιών ή την οργάνωση γενικά των Καραμπινιέρι στην Ιταλία και την, ε, ε, το να επιτρέψει την δημιουργία συνδέσμων. Ε, εάν γίνονται εκλογές μέσα σε αυτά τα σώματα της, της δημόσιας τάξης, οι εκλογές πρέπει να είναι διαφανείς και δημοκρατικές πολλές φορές ζητούν δίκες εκλογές μέσα στα σώματα αυτά, αλλά τους απαντούν με μία... Με σιωπή δεν αντιδρούν καθόλου οι υπεύθυνοι στην κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο κενό οργανωτικό σε αυτό τον τομέα. Ε, εγώ πιστεύω ότι η ενίσχυση αυτών των οργανώσεων ή η τυχόν δημιουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν απειλεί καθόλου το σύστημα. Αλλά άντε να πείσει τους αρμόδιους. Μου φαίνεται ότι ε, ο ρόλος ενός συνδικαλιστή, ο ρόλος ενός μέλους μιας τέτοιας οργάνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικός, πολύ χρήσιμος διότι δείχνει ότι οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι στρατιώτες αισθάνονται ε, μία αξία, ότι τους δίνουμε μία αξία. Εν πάση περιπτώσει τους αναγνωρίζουμε την αξία της ε, δουλειάς τους. Διαφορετικά αποξενώνονται και αποθαρρύνονται. Ε, δυστυχώς στην Ιταλία είμαστε πολύ πίσω στην αναγνώριση της αξίας της εργασίας. Ε, και πιστεύω ότι η δημιουργία τέτοιων ε, στρατιωτικών ενώσεων ε, θα βοηθήσει αυτή την, το έλλειμμα αναγνώρισης. Και η ενεργός συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρουμε τώρα τι κατάσταση επικρατεί στην Ιταλία. Εάν μπορέσουμε να πείσουμε την ιεραρχική αλυσίδα και την κορυφή της ιεραρχίας να μας ακούσει προσεκτικά, κάτι θα επιτύχουμε. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή το προσωπικό εκπροσωπείται σε πάρα πολύ περιορισμένη εμβέλεια, σε πολύ λίγο εκπροσωπείται. Στην παρούσα νομοθεσία 23 μέλη των επιτελείων έγραψαν στον τότε Υπουργό Αλεξάνδρο Περτίνη για τη δημιουργία τέτοιων ενώσεων. Α, όταν διαμορφωνόταν αυτή η νομοθεσία, εννοεί ο μιλητής, έγραψαν μια επιστολή των επιτελείων το 1968 ε, για τη δημιουργία τέτοιων συνδέσμων, αλλά προσέκρουσαν σε ένα τείχος ε, αντίδρασης ε, και δεν έγινε τίποτα τότε. Τότε λοιπόν τους είχαν πει ότι δεν θα αναγνωρίσουμε κανένα τέτοιο δικαίωμα και ούτε κατά διάνοια θα προχωρήσει αυτή η ιδέα. Τώρα όμως έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολλά να κάνουμε. Our... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις προσκεκλημένους μας για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε σήμερα και ελπίζω ότι θα έχω και τη δυνατότητα στο σύντομο χρονικό διάστημα να σας ξαναδώ για το ίδιο για κάποιο άλλο ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα πέντε λεπτών. Until the next session. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας με ένα θέμα που είναι πολύ της ε, μοδός. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μαζί μας τον υποστράτηγο Χόχεν Μπόθ και τον κύριο Βερντιέ από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφοράς, EATC, ε που βρίσκεται στο Εντόβεν κοντά μας λοιπόν. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην δομή αυτή είναι το ότι έχουμε τη δομή αυτή κατά την οποία το pooling and sharing, η συνένωση και η κοινή χρήση είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σαν όρο και έχουμε και την έκθεση του Αντιπροέδρου Λίζεκ της ε, Επιτροπής αυτής που θα ψηφιστεί στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο και αναφέρεται ακριβώς στην εμπειρία αυτή η οποία μας φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα σας ακούσουμε λοιπόν με μεγάλη προσοχή. Η διοικητική αυτή δομή νομίζω ότι υφίσταται εδώ και ένα χρόνο περίπου. Θέλουμε να δούμε ποια είναι τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε, να δούμε πώς δημιουργήθηκε η δομή αυτή Ποιε είναι κατά την άποψή σα ποια είναι τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε και τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και σε άλλου τομεί, πέρα δηλαδή από τι αερομεταφορέ. Ποιε συγκεκριμένε χρήσει μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διοικητική δομής. Πρόκειται λοιπόν για μια δομή την οποία δεν γνωρίζει το ευρύτερο κοινό, δυστυχώ τα έλεγα, αλλά πιστεύω ότι για άλλη μια φορά, δεδομένων των δημοσιονομικών, επιχειρησιακών, λειτουργικών περιορισμών που υπάρχουν ε, στους προπολογισμούς κάθε χώρας ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν δεδομένων όλων αυτών η νέα αυτή διοικητική δομή θα προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών και κυρίως βέβαια των μελών αυτής της Επιτροπής. Κύριε Υποστράτη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω στην ε, Επιτροπή σας στο τέλος του απογεύματος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα θετικά σας λόγια, για αυτά τα οποία μόλις είπατε. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ λίγο στην δική μου την ε, πορεία. Δεν ασχολούμαι ανέκαθεν με τις μεταφορές πιλότος της πολεμικής αεροπορίας και είχα συμμετάσχει σε πολλές επιχειρήσεις διοικητικές στα 39 χρόνια της καριέρας μου, της επαγγελματική μου καριέρας. Ήμουν διοικητής επίσης στην Air Force Academy και επίσης είχα αναλάβει το ρόλο εκπροσώπου πολλές φορές στις σχέσεις που είχαμε με το Υπουργείο Άμυνας και ήμουν επικεφαλής στην ΕΣΔΕΦ για ζητήματα διοίκησης και επίσης ήμουν υπεύθυνο για την αποστολή στο Αφγανιστάν, ιδίω όσον αφορά τις ε, μεταφορές. Εδώ και ένα χρόνο είμαι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Αεροπορικών Μεταφορών, διοίκηση που αποτελεί ένα απτό παράδειγμα του περίφημου pooling and sharing. Είναι παράδειγμα pooling and sharing το οποίο λειτουργεί στην πράξη. Θα ήθελα όμω ε, μαζί σα να σα εξηγήσω για ποιο λόγο το όλο εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα επιτυχέ. Επομένω, είμαι στη διάθεσή σα και για ερωτήσει ή παρατηρήσει μετά την παρέμβασή μου. Πάντω, υπάρχει ένα μοναδικό χαρακτήρα όσον αφορά αυτή τη διοίκηση αεροπορικών μεταφορών. πιστεύω ότι ε, έχει να κάνει με την υποστήριξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής και στρατιωτικής ε, λογικής. Χρειάζονται και οι δύο πτυχές σε αυτή τη διοικητική δομή. Και αν ε, επιθυμεί κανείς να είναι επιτυχή στα πλαίσια πρωτοβουλειών pooling and sharing, συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού πρωτοβουλειών, είναι πολύ σημαντικό να συνδυάζεται η αποτελεσματικότητα μαζί με την αποδοτικότητα της προτινόμενης διοικητικής δομής. Με άλλα λόγια δηλαδή, γνωρίζοντας ότι μειώνονται οι πόροι ακόμα και στον στρατιωτικό κόσμο, ό,τι κερδίσει κανείς σε αποδοτικότητα θα πρέπει να επανεπενδύεται στην κατάρτιση, στην επιμόρφωση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματικότητας, ιδίως όταν πρέπει να ανταποκριθούμε σε πολύ σημαντικές προκλήσεις. Αν καταφέρει κανείς να πετύχει την ισορροπία αυτή, ανάμεσα στην πολιτική και τη στρατιωτική πλευρά και αν καταφέρει να προωθήσει τη δομή αυτή προς την πολιτική πλευρά, τότε ουσιαστικά μπορεί να είναι σίγουρος ότι το όλο εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυχία. Και πιστεύω ότι από γενικής πλευράς μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε δει τελευταία στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αεροπορικών Μεταφορών, βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποιες κέρυες τροποποιήσεις και οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα πλαίσια του ATC, όπου έχουμε τη συμμετοχή χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, οι κάτω χώρες. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε στον εαυτό μας τον απαραίτητο χρόνο, καθώς επίσης και την απαραίτητη βούληση, προκειμένου να προωθήσουμε το βασικό αυτό όραμα. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα ήθελα και εγώ να μοιραστώ τώρα μαζί σας. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ε, σήμερα πιέζονται πάρα πολύ να δείξουν προς τα έξω αυτά αποτελέσματα. Αν δούμε το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Αεροπορικών Μεταφορών, βλέπουμε ότι το όλο εγχείρημα ξεκίνησε στα τέλη του 1990, της δεκαετίας του 1990, όπου αναφερόμασταν σε, κάποια, σε κάποιες νέες στρατηγικές έννοιες, όπου θέλαμε να εξοικονομήσουμε και κάποια χρήματα μετά το, την πτώση του τείχους. Και ήταν δύο οι χώρες αυτές, η Γερμανία και η Γαλλία, που είπαν ότι θέλουμε να επιμεριστούμε τις στρατιωτικές μας ικανότητες όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές και μάλιστα είπαν ε, ότι ε, θέλουμε εν τέλει να παραχωρήσουμε και τμήμα της ε, ηγεσία μας ουσιαστικά και της κυριαρχίας μας, πρέπει να το πω αυτό. Καθορισμένα δηλαδή επίπεδα κυριαρχίας ήταν σε θέση να παραχωρήσουν αυτές οι δύο χώρες και στη συνέχεια περνάμε σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θίξετε κι εσείς κύριε Πρόεδρε, τις διάφορες πρωτοβουλίες συνένωσης και κοινή χρήση που έχουμε επιτάπητος εδώ και ένα χρόνο και προφανώς ένα παράδειγμα pooling and sharing αποτελεί η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αεροπορικών Μεταφορών. Προσπαθούμε μέσω του EATC να ανταποκριθούμε στις, στη γενικότερη τάση μείωση των πόρων και να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στο επίπεδο φιλοδοξίας της πολιτική ηγεσία μας, καθώς επίσης και της δέσμευση της στρατιωτική που θα θέλαμε να πετύχουμε στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προσέγγισης. και κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι νέο, αλλά πρέπει να τονίσουμε. Έχουμε και την πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Γκέιτς, ο πρώην υπουργό Άμυνα, ήρθε στις Βρυξέλλες και μίλησε για το Smart Defense Initiative. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Διοίκηση αεροπαρικών Μεταφορών αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα του, της Ευρωπαϊκής ε, Συνεργασίας, όπου έχουμε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταφέρουν να συνεργαστούν αποτελεσματικά στα πλαίσια ενός ε, επιτυχούς εγχειρήματο. Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αεροπερικών Μεταφορών έχει επιχειρήσεις υποστήριξης και έχει δυνατότητες και, στις, και στους δύο τομείς. Όσον αφορά τον τομέα pooling, της εκμετάλλευσης, της συνένωσης, προσπαθούμε να συγκεράσουμε όλους τους πόρους που έχουμε από όλε τις διαφορετικές δομές και σας, θα σας δείξω υπό τη διοίκησή μου για πόσους πόρους μιλάμε και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις, όλους πόρους σε ένα κεντρικό σημείο όπου υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα διοίκησης. Καταφέρνουμε κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε συνέργειες και καταφέρουμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Αυτό όσον αφορά την εκμετάλλευση. Περνάμε πίτα στον τομέα του επιμερισμού, του sharing. Προσπαθούμε να επιμερίσουμε τις ικανότητες, τις δυνατότητες αυτές σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στις διάφορες επιχειρήσεις ε, ιατρικής ε, και Βλέπουμε λοιπόν στην πράξη ότι έχουμε μια συνεργασία μεταξύ χωρών όπως η ε, Γερμανία, η Γαλλία, οι κάτω χώρες που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένε ανάγκες των χωρών αυτών και ουσιαστικά οι χώρες αυτές, χάρη στην, ε, τον των, των ικανοτήτων, δεν χρειάζεται να αγοράσουν ακριβές πλατφόρμες και δεν χρειάζεται επίσης να καταφύγουν στην εξωτερική ανάθεση των επιχειρήσεων αυτών. Προσπαθούμε να καταφέρουμε να συντονίσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες μεταφοράς στρατιωτικών εμπαρευμάτων. Δεν μπορούμε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε ότι θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Θέτουμε συγκεκριμένε φιλοδοξίες και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές. Βλέπουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να δεσμευτούμε και σε ποιους τομείς μπορούμε να επενδύσουμε τις στρατιωτικές μας δυνατότητες. Είναι πολύ σημαντικό σαφώς να λαμβάνουμε υπόψη μας την, μείωση, των στρατιωτικών πόρων και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα οποιασδήποτε εξοικονόμησης επιτυγχάνεται να επενδύουμε σε τομείς όπου χρειάζεται να έχουμε μεγαλύτερη παρουσία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες προσπαθούν να επενδύσουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν θα έχω εγώ τον απόλυτο έλεγχο βέβαια των στρατικών αυτών δυνατοτήτων που έχουμε συγκεκριμένε περιοχέ. Αυτό γίνεται από ευρωπαϊκέ δομέ διοίκηση ελέγχου έκτακτη ανάγκη. Και βέβαια κάθε χώρα πρέπει να παραχωρήσει και κάτι. Το χειρότερο βέβαια για κάθε χώρα είναι να παραχωρήσει μέρος της κυριαρχίας της. Εν τέλει πάντως πρέπει να καταλήξουμε σε, πολύ, σε μια πολύ ευφύ Έννοια, είναι ένα πολύ ευφυέ εγχείρημα και θα σας δείξω τελικά πώ η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αεροπορικών Μεταφορών μπορεί να λειτουργήσει προ προς αυτό. Δηλαδή να έχουμε μία έξυπνη προσέγγιση όπου ε, οι χώρες ε, καταφέρουν να κερδίσουν σε αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα μέσω μικρών παραχωρήσεων. Μία ομάδα η οποία δημιουργήθηκε Ε, με τον προκάτοχο του, e, EATC. Ξεκινήσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία, γαλλογερμανική-ολλανδική πρωτοβουλία και έχουμε φτάσει μέχρι το 2010 που δημιουργήθηκε τελικά η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αεροπορικών Μεταφορών. Είχαμε κάποιες, ενδιάμος, ενδιά, κάποιες ενδιάμεσες δομές. Είχαμε την ε, Ευρωπαϊκή Δομή Αερομεταφορών στο Ενχόφεν και αυτή Προσπαθούσαμε να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και ιστορικά οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν έναν τομέα στον οποίο προσπαθούν οι χώρες να συνεργαστούν όλο και περισσότερο. Και εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό μέσω του pooling and sharing. Πάντως κάθε φορά που επικεντρωνόμαστε σε κάποιες ιστορικές κοινέ συνεργασίες κάθε φορά προσπαθούμε να εντοπίσουμε τομεί συνεργασία, βρισκόμαστε και στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Από στρατιωτικής ε, πλευράς είναι εύκολο να μιλάει κανείς για στρατιωτικές επιχειρήσει, όπου έχουμε ε, κεντρικό έλεγχο, κεντρική διοίκηση και έναν ε, επικεφαλής και άλλο πράγμα βέβαια είναι οι πιο αποκεντρωμένες ε, επιχειρήσεις. Αυτό είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα στο οποίο ήθελα να αναφερθώ και από την άλλη ήθελα να σας πω και το ακόλουθο. Στα πλαίσια των αεροπορικών μεταφορών αναφερόμαστε επίσης και στην, στον εντοπισμό μιας συγκεκριμένη νοοτροπίας κοινή εργασίας. Γάλλοι, Γερμανοί, οι δήμονες στα πλαίσια των αεροπορικών μεταφορών πρέπει να συνεργαστούν και αυτό κάνανε στην Αφρική ε, για να αντιμετωπίσουν διάφορα φαινόμενα, για να αντιμετωπίσουν φυσικές καταστροφές. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του τσουνάμι. Επίσης, ε, έχουμε μια μακρά ιστορία στο να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση κοινών πρακτικών. Αν ένας Βέλγος αλεξιτοπτιστής ε, πρέπει να εργαστεί στα πλαίσια μιας κοινή δράσης, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Ενδεχομένω ένας διοικητή να μας πει ότι η άδεια για αυτό το αεροσκάφο δεν είναι δική σα ευθύνη. Κατά τη διάρκεια τέτοιων κοινών επιχειρήσεων είχαμε περιπτώσεις ότι, όπου κάποια αεροσκάφη έπρεπε να επιστρέψουν στη βάση τους γιατί ε, είχαν ε, εξοπλιστεί τα αεροσκάφη αυτά με εντελώ διαφορετικό τρόπο από αυτόν προβλεπόταν από τον γερμανικό στρατό. ότι υπάρχουν λοιπόν κάποια κοινά μέτρα αδειοδότησης... πρέπει να καταλήξουμε και σε κάποιου κοινούς κανονισμούς... κοινέ τεχνικές και κοινέ διαδικασίες... προκειμένου να μην μειωθεί η αποτελεσματικότητά μα. Στα πλαίσια λοιπόν του EATC, τα κράτη αποφάσισαν σιγά σιγά να μεταφέρουν όλες αυτές τις εθνικές ευθύνες, καθώς επίσης ε, και την ευθύνη και την αρμοδιότητα που υπάρχει για την επιτήρηση του ε, ελέγχου. Και μετέφεραν επίσης ε, όλη αυτή την κοινή προσέγγιση όσον αφορά ένα κοινό στρατοτικό όραμα, τα κοινά στρατοτικά δόγματα. Όλες αυτές οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην ενιαία Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αεροπορικών Μεταφορών. Ο τελικός στόχος ήταν να καταφέρουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί και να καταφέρουμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των υφιστάμενων πόρων. Προκειμένου όμως να πετύχουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να καταλήξουμε σε έναν ευφυή σχεδιασμό σε αυτόν ακριβώς κατέληξε μια ομάδα μετά από μια σκληρή εργασία δύο ετών και μετά από μια συγκεκριμένη εντολή που τους δόθηκε. Άρχισε να εργάζονται το 2006, στις αρχές του 2006 και δύο χρόνια μετά το Βέλγιο, οι κάτω χώρες, η Γερμανία και η Γαλλία κατάφεραν να καταλήξουν στην στρατηγική αυτή έννοια του ATC, την οποία βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε δύο αλληλοεξαρτώμενους πυλώνες, και βασικό στοιχείο εδώ πέρα είναι ότι προβλέπεται μία ελεγχόμενη παραχώρηση, παραχώρηση ενό ενός τμήματος της κυριαρχίας. Ουσιαστικά, τα κράτη-μέλη παραθέτουν εδώ πέρα ένα μεγάλο βαθμό διαθεσιμότητας του ενεργητικού τους, των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων και αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του συστήματος. Ουσιαστικά προϋποθέτει αυτή την υποόρους παραχώρηση της κυριαρχίας. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν σε ποιο βαθμό θα κάνουν την παραχώρηση αυτή. Και τα κράτη-μέλη ανα πάσα στιγμή μπορούν να ανακαλέσουν ή να καταργήσουν αυτή τη μεταφορά ηγεσία. Βέβαια, αν υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο εμπιστοσύνη, αν υπάρχουν τα κατάλληλε συνθήκε συνεργασία, δεν πρόκειται τα κράτη-μέλη να επανέλθουν να αναθεωρήσουν αυτή την παραχώρηση κυριαρχία. Όσον αφορά τώρα το λειτουργικό πυλώνα, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να κατακαιρματίσουν τον λειτουργικό αυτόν τομέα σε κάποιους υποτομείς και προβλέπεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο ηγεσία για τον καθέναν από τους υποτομείς αυτούς. Για παράδειγμα, εγώ έχω την διοικητική ηγεσία όσον αφορά τη σύνταξη των εγγράφων και όσον αφορά τις ε, αεροπορικές ε, μεταφορές της ε, γερμανικής αεροπορίας για τα προγράμματα κατάρτισης. Εγώ ουσιαστικά καθορίζω τι θα πρέπει να πετύχει η γερμανική πολεμική αεροπορία στους συγκεκριμένου στόχους που θέτουμε. Είμαι επικεφαλής όμως διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης και είμαι σε θέση επίσης να έχω μια διοικητική θέση και για, τις υπόλοιπες, και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια χώρα η οποία μπορεί τουλάχιστον να είναι επικεφαλής αυτής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Αεροπορικών Μεταφορών. Είμαι σε θέση κατά αυτόν τον τρόπο να δω ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικέ και είμαι σε θέση να ενσωματώσω, για παράδειγμα, τι γαλλικέ προοπτικέ σε συγκεκριμένου τομεί δράση. Και εν τέλει, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κράτη τα οποία είναι σε θέση να ακολουθήσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Ας περάσουμε στη διαφάνεια της εμπιστοσύνης ε, και της αυτοπεποίθησης. Βλέπετε ότι η πλειοψηφία των αεροσκαφών ε, χρησιμοποιούνται από τη δική μας διοίκηση και σαφέστατα από εθνικής πλευράς υπάρχει ε, αυτή η βούληση εκχώρησης ε, κυριαρχίας ε, λόγω των φιλοδοξιών που υπάρχουν. Η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, πρόεδρε, το γνωρίζετε κι εσείς ότι ε χρειάζονται, χρειάζεται προσωπικό, έχετε ειδικά αεροσκάφη, χρειάζεται υποστήριξη επιχειρήσεων φυσικά δεν ζητώ εγώ την διοίκηση αυτών των πόρων. Η Γαλλία ε, κρατά την εξουσία που έχει σε σχέση με τα αεροσκάφη εν συγκρίση με την ε, Γερμανία. Ε, είναι σαφές ότι τα γερμανικά αεροσκάφη παραμένουν υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Τα το, ο αεροσκάφος 340 της ε, κυρίας Μέρκελ που χρησιμοποιείται για ε, ε, κρατικές πτήσεις, για πτήσεις των βουλευτών. Φυσικά υπάγονται στην ίδια διοίκηση. Ε, ακόμη και εκεί έχουμε ε, διαρκή μείωση των πόρων Ακόμη και για τα τακτικά αεροσκάφη, οι Γερμανοί κάνουν περικοπές σε σχέση με τα 360, οι Γάλλοι εταίροι τους το ίδιο κάνουν. Έχουμε αρχίσει αναθεώρηση του στόλου, δηλαδή συνδυασμένη προσέγγιση για να δούμε πώς η σταδιακή μείωση των πόρων μπορεί να συνδυαστεί ε, με διατήρηση των ικανοτήτων μας και αύξηση αυτών. Ε, και αυτά σε συνδυασμό με την θέση σε ισχύ του, της νέας γενιάς αεροσκαφών. Επόμενη διαφάνεια, τα επιτεύγματα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε καταλήξει σε ε, διάφορες πολύ σημαντικές αλλαγές που έχουν σημειώσει επιτυχία και ε, παρέχουμε κυρίως αυτές τις δυνατότητες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Η διοίκηση αυτή δεν ε, λειτουργεί εκ παραλίλου με διάφορες περιφερειακές ευρωπαϊκές οργανώσεις. Εμείς συνδεόμαστε πολύ στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Έχουμε αναπτύξει μια σχετικά καλή συνδεσιμότητα των στόλων. Έχουμε επίσης στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό ε, Όμιλο ε, για τις αερομεταφορές. Τώρα, κοινή ε, διπλωματική άδεια. Όταν υπάρχει κοινό ενδιαφέρον ε, για την ε, μέθοδό μας, ζητείται αυτή η κοινή άδεια. Δηλαδή, η κοινή άδεια επιτρέπει χωρίς επιπρόσθετη άδεια να μεταφέρει κάποιος απευθείας από τη Γερμανία στην Ογλεά, στη Γαλλία, ένα επικίνδυνο φορτίο παραδείγματος χάρη. Δεν χρειάζεται ε, παρά μόνο η πρώτερη έγκριση των κρατών να μετάσχουν σε αυτόν τον σχηματισμό. Τώρα, σε σχέση με τα πληρώματα και την αρμόνιση της, ε, ε, των κανονισμών σε σχέση με τα πληρώματα. Στο Κονγκό δημιουργεί, είχαμε μια ιδιαίτερα επιτυχή ευρωπαϊκή αποστολή και όχι μόνο αντιμετωπίστηκε το θέμα της ε, διεθνικής, ε, διεθνικού προσδιορισμού καθηκόντων, όχι μόνο χρησιμοποίησαμε από κοινού αεροσκάφη, το πρόβλημα ήταν ε, να εντοπίσουμε τα διάφορα επίπεδα του πληρώματος. Δεν υπήρχε γενική επισκόπηση των ικανοτήτων ως προς το πλήρωμα, γιατί κάποιοι μπορούσαν να πετούν μόνο για 12 ώρες, άλλοι για 16, οπότε για την ανάπτυξη ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί για το προσωπικό και άρα χρειάζεται μια πιστοποίηση για να καταλήξουμε σε εναρμόνιση και πιστεύω ότι ε, έχουμε καταφέρει να εναρμονίσουμε την προσέγγιση των τεσσάρων αυτών ε, κρατών που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία. Σχετικά με την ιατρική τεχνογνωσία και την ιατρική εκένωση, αναφέρθηκα σε αυτό, ε, προκύπτει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων ε, και επ' αυτού συνεργαζόμαστε στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Άμυνα. Επιπροσθέτω, κάνουμε μια, ένα πιο συνετό στρατιωτικό ε, σχεδιασμό. Όταν μιλάμε για την παρατήρηση των, των εκλογών που γίνονται τώρα στο Κονγκό, εξετάζουμε ποιοι είναι οι πόροι που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε σε αυτό το κράτος ε, διότι δεν ε, έχει, ε, σε περίπτωση μάλλον που επιγόντως θα πρέπει να αποχωρήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και δεν υπάρχει προς το παρόν αντίστοιχη δομή. Από καταλαβαίνετε όμως μια τέτοια επιχείρηση προϋποθέτει πολιτική εντολή. Ε, στη συνέχεια ο πίνακας ε, επιδόσεων, έτσι θα τον αποκαλέσω. Ε, μεγάλη επιτυχία, ομολογουμένως. Ε, δεν κρύβονται αποτυχίες και καταγγελίες πίσω από τον πίνακα. γράφεται μια ιστορία ουσιαστικά και χτυπάω ξύλο. Ε, διότι οι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτε υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δράση της Ευρωπαϊκής Διοίκηση Αερομεταφορών. Ε, θα σχολιάσω και πάλι το τμήμα με για ε, ε, την μεταφορά τραυματιών ε, δηλαδή για τη πτήσεις υγειονομική εκένωση. Βλέπετε ότι εκεί σημειώνεται η μεγαλύτερη επιτυχία. Δεν χρειάζεται τώρα να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το 2010... Όταν ε, αρχίσαμε είχαμε περίπου 600 ώρες ε, διεθνικών πτήσεων. Ε, τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Γερμανοί ευρωβουλευτές να μπουν ας πούμε σε ένα αεροσκάφο. Έγινε και αυτό ε, στο Κολόμπο για να πάνε στην σύσκεψη ε, Υπουργών ε, Άμυνας για τις νέε δομέ των ενοπλέων δυνάμεων. Ένα βελγικό 130 πήρε όλους τους υπουργούς και τους πήγε στο Βερολίνο. Βλέπετε τα ωφέλη της κοινή μεταφοράς υποστηρίζονται και επιχειρήσεις όπως η ΆΙΖΑΦ αλλά και άλλες. Είδου οι επιτυχίες ε, που έχουμε καταγράψει και άρα πραγματικά έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας. Επόμενη διαφάνεια, ε, περί τίνος πρόκειται, επιχειρησιακό όφελος. Δεν χρειάζεται όμως να δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια έχουμε με, συμμετάσχει σε κοινέ ε, ε, πτήσεις προστασίας. Ε, ε παραδείγματος χάρη, οι προσπάθειες που γίνονταν από τι γαλλικέ δυνάμεις αντικαταστάθηκαν από τι κοινέ δυνάμεις. Ε, Παραδείγματο χάρη έφυγαν δυνάμεις από τη Βόρεια Γαλλία για να υποστηρίξουν ε, τις ε, ένοπλες δυνάμεις στο Νότο. Είναι θέμα χρονισμού επίσης όταν χρειάζεται κοινή τέτοια πτήση. Ε, παρατηρούμε πολλά ωφέλη, έλαβα και σχετικές επιστολές και ε, οι, 20% των υποστηρικτικών επτήσεων για τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ε, γινόταν με αεροσκάφη από το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αναφέρω χαρακτηριστικά. Επόμενη διαφάνεια είναι οι τρεις τελευταίες διαφάνειες και θα ήθελα να σας ε, μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφοράς ε, είναι ένα σχέδιο, θα έλεγα, για μια μελλοντική ε, πολιτική συνεκμετάλλευσης και επιμερισμού. Πιστεύω ότι έχουμε βελτιωθεί ως προς τη βελτιστοποίηση της χρήσης των μέσων. Μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση ε, ή να επενδύσουμε σε αυτές ε, τις ε, ε τις κοινέ πτήσεις. Reduction of overhead cost. Don't please. Σε σχέση με τη μείωση του κόστους, Υπάρχουν πολλοί τομεί όπου έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση. Παραδείγματο χάρη κάνουμε εξωτερική ανάθεση για την Ολλανδική Ιατρική Εκένωση. Επίσης ο σχεδιασμός ε, γίνεται πολύ πιο οικονομικός ε, με την κοινή χρήση των ε, μέσων. Επίσης δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη λογιστική, υλικοτεχνική υποστήριξη πλέον για αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Ποιες είναι οι προκλήσεις. Πιστεύουμε ότι ανοίγουμε σε αυτή τη δομή των τεσσάρων κρατών και είναι σχετικά σημαντική αυτή η δήλωση όταν ε, ε, ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μου είπανε καλωσορίσατε αλλά πλέον δεν είστε Γάλλος ε, στρατηγός και ο συνάδελφός μου που κάθεται στα αριστερά μου αυτό μου είπε, δηλαδή είμαστε πλέον διεθνικοί διότι διασχίζουμε τις συνοριακές γραμμές όλων των ενόπλων δυνάμεων σε αυτές τις τέσσερις χώρες χάρη στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφοράς. Αν τώρα αυξήσουμε ε, και τον αριθμό των μελών θα έχουμε ε, πετύχει το στόχο μας. Ε, φυσικά δεν είναι αυτονόητο να συνειδητοποιήσουν ότι το επιτελείο των οπλικών συστημάτων της Γερμανίας έχει σε ένα ορισμένο βαθμό ενταχθεί σε αυτή την κοινή δομή. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με την οτροπία και την φράσεολογία, ε, ε, μάλλον ε, το γλωσσικό ζήτημα. Ε, δεν ε, ομιλούν όλοι την αγγλική, δεν είναι η αγγλική μητρική γλώσσα όλων. Για την αεροπορία τα αγγλικά είναι η κοινή γλώσσα, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα ε, σετ επισήμων γλώσσα. Μην ξεχνάτε ότι όλοι θα πρέπει να μιλάνε αγγλικά. Ε, και όχι μόνο να μιλάνε αλλά και να έχουν τα έγγραφα στα αγγλικά για την πρόσληψη του προσωπικού που συνήθως είναι στα γαλλικά ή στα γερμανικά συνεχώ πρέπει να μεταφράζονται προς τα αγγλικά γιατί αλλιώς δεν προβλέπεται συμμετοχή σε αυτή την ε, πολυεθνική δομή μόνο έτσι μπορούν να λειτουργήσουν οι κοινέ ε, στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις. Ε, ούτως ή άλλως έτσι λειτουργεί οποιοδήποτε διεθνικός οργανισμός, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει διαφάνεια. Κοινωνικές επιτυχίες από την πλευρά μας, θα έλεγα για τις προκλήσεις ότι το Eindhoven είναι μια θεσπέσια πόλη συγχαίρω τους ε, Ολλανδούς συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ ωραία η πόλη για την ε, ε, παιδεία, τη σχολική εκπαίδευση. Θα ζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ειδική πρόβλεψη για τους λίγους μαθητές που έχουμε, διότι στο Άιντχόφεν δεν υπάρχει διδασκαλία για την απόκτηση του ευρωπαϊκού ε, απολυτηρίου και θα ζητήσουμε την ένταξη των μαθητών στα ευρωπαϊκά σχολεία. Ελπίζουμε να μας υποστηρίξετε. Για... Ως προς τις επιχειρησιακές ικανότητες Νομίζω ότι μέχρι το 2012 θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και το θέμα της προσχώρησης του Λουξεμβούργου στη δομή είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Ε, στην επόμενη ε, συνεδρίαση των επιθεωρητών θα προσκαλέσουμε τον εκπρόσωπο της χώρας ε, ευελπιστούμε ότι το 2013 και 2014 θα έχουμε ολοκληρώσει το νομικό πλαίσιο για την προσχώρηση νέων ε, ε μελών. Στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ε, τώρα, αν ε, πρόκειται για πρότυπο αυτή η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφορές σχετικά με τη συνεκμετάλλευση, ε, είναι πολύ διάζουσα η δομή ε, της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Αερομεταφορών. Ε, προσπάθησα να στο, στο μεταφέρω. Παράπλευρες απόλυτες πάντως δεν μπορούν να αποδοθούν στη δική μας διοίκηση. Δεν σκοτώνουμε ανθρώπους. 90% των επιχειρήσεων βασίζονται στην υποστήριξη. αυτό που χρειάζεται επίσης είναι να παραμένουν διαθέσιμε οι χώρες που μετέχουν σε αυτή τη δομή. Όταν ε, κανείς ε, προσπαθεί να καταλήξει σε μία νέα ευφύ τέτοια στρατηγική έννοια, Νομίζω ότι μπορεί να αποκομίσει κάποια πολύ χρήσιμα διδάγματα από τη δική μας εμπειρία για την συνεκμετάλλευση και τον ε, επιμερισμό. Από πλευράς μου θα έλεγα ότι ένα ή δύο κράτη θα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα και να παραχωρήσουν κάτι, να υποχωρήσουν. Δεν, ε, ε, όχι απαραίτητα την κυριαρχία τους, αλλά να κάνουν μια προσπάθεια. Τώρα, στρατιωτική προστιθέμενη αξία. Άλλο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα κατά τη γνώμη μου. Ε, Ε, θα χρειαστεί επίσης οι εθνικοί στόχοι να περιοριστούν προς όφελος των διεθνικών. Επίσης, σας είπα ότι χρειάζεται ευφυή σχεδιασμός και ε, συγκεκριμένη εντολή. Ε, κατόπιν συγκερασμός των ε, διαφορετικών ε, νοοτροπιών και να λυθεί το γλωσσικό ε, πρόβλημα και να υποστηρίξουμε το γενικότερο όραμα, αν θέλετε, αυτή της κοινή δομή. Euh, euh, Ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη αυτή δυναμική παρουσίαση, η οποία επέμεινε σε όλα τα σημαντικά σημεία αλλά και σε αυτά τα οποία θα μπορούσαν ακόμα να εξελιχθούν περισσότερο στα πλαίσια της δομής αυτής. Νομίζω ότι ε, πολύ εξημών ανακαλύψαμε την ε, διοικητική αυτή δομή για πρώτη φορά σήμερα. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση. Ήσασταν ιδιαίτερα πλήρης, διεξοδικός. Δεν έχω ερωτήματα να σας θέσω. Αναρωτιόμουν μόνο για τη δυνατότητα διεύρυνσης της διοικητικής αυτής δομής. Συναφερθήκατε στο Λουξεμβούργο. Έχουν εκδηλώσει και άλλες χώρες ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αεροπορικών Μεταφορών και κατά την άποψή σας ποιες είναι οι πιθανές υποψήφιες χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση EATC. και ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι χώρες αυτές προκειμένου να ενταχθούν. Είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα, είναι και ζήτημα ικανοτήτων, υλικών ικανοτήτων ή όσον αφορά το ανθρώπινο προσωπικό. Είναι ένα συνδυασμό όλων αυτών τελικά. Ή τελικά πρόκειται για μια καθαρά πολιτική απόφαση για το αν θα ενταχθεί ή όχι μια χώρα στην EATC και σας έχουν προσεγγίσει για το ζήτημα αυτό, για τη διεύρυνση δηλαδή του EATC. Πολλοί θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στον Αντιπρόεδρο Λίζεκ, ο οποίος συνέταξε και την έκθεσή μας, η οποία αναφέρεται στο pooling and sharing. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας χειροκροτήσω θερμά, κύριε υποστράτη, γιατί δείξατε ξεκάθαρα σήμερα ότι αυτά που αναφέρω στο σχέδιο γνωμοδότησης είναι ακριβώς αυτά τα οποία υποστηρίζετε. Είναι πάρα πολύ σωστές οι σκέψεις σας και χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα αυτά που είπατε, διότι επιβεβαιώνουν τη δική μας κοινή θέση και τις δικές μας απόψεις που παρουσιάζονται στο σχέδιο γνωμοδότησης. Για να σας ενημερώσω, κύριε Υποστράτη, κάνουμε και ορισμένα όνειρα στην έκθεσή μας. Αυτό το ο επιμερισμός ε, και ο, η συνεκμετάλλευση είναι ένας επιθυμητός στόχος όλων μας. Και έχω και μία ερώτηση προς εσάς, αλλά βασικά είναι πολιτική φύσεως. Στην Πολωνία λέμε, εάν τα πράγματα βαίνουν καλώς, γιατί η κατάσταση διαγράφεται τόσο κακή. Ε, δεν ε, θα ρωτήσω βεβαίως γιατί η Πολωνία δεν ανήκει στην Ένωση Αερομεταφορών. Αυτό πρέπει το ερώτημα να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό στην Πολωνία και να απαντήσει εκείνος. Όμως ε, θα ήθελα να ξέρω από εσά. Η Ιταλία, η Ισπανία που έχουν μεγάλο πολιτικό δυναμικό μπορούν ε, να συμμετάσχουν και μπορούν να φέρουν, να επιφέρουν ένα μεγάλο όφελος. Συμμετέχουν ή όχι και αν όχι σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκάιλερ, και εγώ ευχαριστώ για αυτήν την ολοκληρωμένη παρουσίαση και με, ενθουσιάζει το γεγονός για το πόσο ωραία μπορεί να μιλήσει για τις αερομεταφορές ένας πιλότος αεροπλάνων jet διότι η εργασία είναι ευχαρίστηση με αυτές τις συνθήκες. Θα ήθελα ε, να σήξω ορισμένα σημεία που με ενδιαφέρουν. Ε, λέει ότι ο στόχος της EATC είναι να ε, προσχωρήσουν όλες οι εθνικές αρμοδιότητες προς την EATC των διασυνοριακών αερομεταφορών. Από απόψεως διαδικασιών τώρα, πού βρισκόμαστε και τι μεταφορά κυριαρχίας έχει επέλθει μέχρι τώρα. Μήπως ε, θα πρέπει όλες αυτές οι αρμοδιότητες να συγκεραστούν ε, υπό την EATC και αναφέρεται εδώ σε αεροσκάφη με σταθερά πτερίγια. Δεν καλύπτει δηλαδή τα ελικόπτερα ή έτσι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Εν συνεχεία ε, υπάρχουν ε, μνημόνια συνεργασίας. Αυτή είναι η βάση δηλαδή ε, της συνεργασίας μας. Τώρα όμως έχουμε καινούργιες συμβατικές διαδικασίες που είναι δεσμευτικές. Και σκέφτομαι μήπως μπορούμε να υπερβούμε αυτά τα μνημόνια και να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα πλαίσιο δομημένης συνεργασίας, structured cooperation, έτσι ώστε να υπάρχει και μια συμβατική δομή, μια συμβατική, ένα ε, συμβατικό πλαίσιο στη συνεργασία αυτή. Επίσης, πώς διαμορφώνεται η συνεργασία σας με, αυτήν την ενδιάμεση, με το ενδιάμεσο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ. Επίσης αναφέρατε και την ε, την υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας ότι αυτή διαχειρίζεται τον Ευρωπαϊκό Στόλο Αερομεταφορών και ότι είναι συναρμόδια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης. Μήπως θα μπορούσατε εσείς να λάβετε αυτό το, την πτυχή της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Ε, ας πούμε ε, σεμινάρια ε, ή ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τις αερομεταφορές εκένωσης, ιατρικές ή άλλου είδους. Η Γερμανία έχει μία εθνική διοίκηση η οποία ενσωματώθηκε σε εσά. Τι γίνεται όμως αν υπάρχει μια άλλη εθνική διοίκηση η οποία δεν υπάρχει στην ATC ε, και πάλι και αναφέρεται σε αερομεταφορές. Ε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, εγώ χωριστά. Ευχαριστώ ο κύριος Κάμπελ Μπάρονμαν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ποστάτη για την ε, παρουσίασή σας. Έχω δύο ερωτήματα. Καταρχάς αναφέρεται στο άρθρο στην έκθεσή σας ότι αυτή τη στιγμή συντελείται ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό εννοούμε με συνεκμετάλλευση και επιμερισμό. Εννοούμε στρατιωτική ολοκλήρωση, ενσωμάτωση, δηλαδή η δημιουργία μιας ε, στρατιωτικής Ευρώπης. Αυτή την κατεύθυνση επισημούμε ή προστακυβαίνουμε. Η δεύτερη ερώτηση και πάλι στην έκθεση αναφέρεται ότι αρχικά το ΝΑΤΟ είχε ε, εξουσιοδιωτήσει αυτή τις ε, διαδικασίες. Γιατί δεν πέρασε όλη αυτή η επιχείρηση αερομεταφρών από το ΝΑΤΟ και έγινε ένας ξεχωριστός φορέας. Υπάρχουν διαφορετικές, ε, ένα διαφορετικό δυναμικό και μια διαφορετική, διαφορετικές Δυνάμει που ενεργούν και αποδοτικότητες οι οποίε πρέπει να λάβουμε υπόψη που δεν μπορεί να περάσουν από το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να απαντήσω κατά σειρά τις ερωτήσεις. Αρχίζω με, την... με το ερώτημα για τη διεύρυνση της υπηρεσίας μας, της διοίκησής μας σχεδιάζοντας ε, την διοίκηση αυτή επί τη βάση τεσσάρων κρατών, δηλώσαμε ότι είμαστε μια ανοιχτή, ανοιχτή, ένας ανοιχτός φορέας. Ε, ε, βεβαίως, βάσει πολιτικών αποφάσεων, πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς τις δομές και να εφαρμόσουμε την κατάλληλη διαδικασία για να προσχωρήσουν και άλλα κράτη. Αυτό ακριβώς θα γίνει με το Λουξεμβούργο. Τώρα γιατί το Λουξεμβούργο είναι το πρώτο κράτος που θα προσχωρήσει. Ε, αυτή είναι η κατάλληλη συνέχιση των διαδικασιών ευρωπαϊκού συντονισμού. Έχουμε βρετανικές, νορβηγικές, εξ, λουξεμβουριανές ε, πτυχές και όταν το 2006 έγιναν οι πρώτες ενέργειες από την Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, το Βέλγιο ήταν κάπως επιφυλακτικό. Είπε όμως ότι ε, ε, στο τέλος της ημέρας θέλουν να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση Μεταφοράς. Είναι λοιπόν μια ειδική περίπτωση του Λουξεμβούργου. Ναι, μεν δεν μπήκε στην αρχή, αλλά θα μπει τώρα. Και ε, για το ερώτημα λοιπόν της διεύρυνσης, εδώ θα δώσω και αν θα πρέπει η αεροπορία να συμμετάσχει, θα δώσω την ίδια απάντηση. Ένα κράτος το οποίο θέλει να χρησιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφοράς για να διευρύνει το δυναμικό και την αποτελεσματικότητά του μπορεί να, ε, πρέπει μάλλον να συμμορφώνεται με ορισμένα κριτήρια. Θα πρέπει να προσδίδει στρατιωτική προστιθέμενη αξία. Ε, δεν ισχύει κυριολεκτικά αυτό, αλλά γενικά ως προσέγγιση πρέπει να προσφέρει κάτι από απόψεως ε, στατιωτικής ε, αποδοτικότητας. Υπάρχουν ορισμένες διαθροτικές στρατηγικές προϋποθέσεις που πρέπει να γίνουν σεβαστές. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το θέμα του κόστους. Εάν οι Γερμανοί πετούν για να υποστηρίξουν γαλλικές επιχειρήσεις στο Χάρματαν, Αυτές οι πτήσεις ε, πρέπει να εξισορροπηθούν και από απόψεως κόστους, δαπανών δηλαδή. Ε, πρέπει να προσέξουμε την οικονομική δαπάνη να επιμερίζεται μεταξύ των ε, κρατών. Δεν μπορεί ένα κράτος να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ή μονομερό το δυναμικό ενός άλλου κράτους χωρίς να υπάρχει μια αντιστάθμιση. Επίσης ε, πρέπει να συνυπογράψει τη συνθήκη. Και εσείς ως μέλη του Κοινοβουλίου το ξέρετε αυτό πολύ καλά και μπορείτε να το προωθήσετε. Αυτή τη στιγμή το EATC δεν βασίζεται σε μνημόνιο. So, what is that? I'm, uh, very much... Μνημόνιο αλλά θέλουμε να βασίζεται σε συμβατικές υποχρεώσεις. Αυτό αφορά ιδιαίτερα και τη διαδικασία προμηθειών, procurements. Μην ξεχνάτε και την τεχνολογία πληροφορικής, IT connectivity. Αν εγώ θέλω να έχω το πλεονέκτημα ε, της προμήθειας ε, τεχνολογίες πληροφορικής ε, με τα χρήματα των φορολογούμενων αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω τις προημήσεις με την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών της Ολλανδίας και με καλύπτει. Είμαι λοιπόν εγώ υπόλογος σε μια οργάνωση ομπρέλα, σε μια οργάνωση που επικαλύπτει ε, διασυνοριακά τις αρμοδιότητες και σε άλλα θέματα, εργατικά, διοικητικά. Ε, επειδή είμαστε μια διασυνοριακή και διακρατική οργάνωση, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτή τη συνθήκη, αυτή τη την, ε, της βάση, ε, τη θεσμική βάση λειτουργίας. Είμαστε μια μόνιμη δομή. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ενέργειας και συγκεκριμένο πεδίο ισχύω για τις αρμοδιότητές μας χωρίς αμφισβητήσεις και ε, δεδομένου ότι ε, συνεργαζόμαστε εκτός των τεσσάρων αυτών ιδρυτικών ε, κρατών και με άλλα κράτη σε κοινέ επιχειρήσεις πρέπει να έχουμε ένα εξαιρετικά σαφές θεσμικό πλαίσιο. Εφόσον λοιπόν συνυπογράψουν το καταστατικό λειτουργία, συνθήκη λειτουργία, θα πρέπει να συμμετάσχουν και στον κοινό προπολογισμό. και εκεί ακριβώς θα κρυθεί ποια θα είναι συμβολή ενός κράτους μέλους στην EATC. Εάν θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει το δυναμικό, το γερμανικό δυναμικό, θα πρέπει να συμβάλλει, ε, να προσφέρει ας πούμε προσωπικό, να προσφέρει ανθρώπινο δυναμικό, που θα βοηθήσει στην επιχείρηση. Επίσης, δεν θα δεν ε, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, το κοινό, τα κοινά συστήματα πληροφορικής τα οποία είναι ορατά και προσβάσιμα από 400 άλλους πελάτες. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να υπάρχει μία κοινή ε, βάση χρήσης αυτής της ευρείας βάσης πληροφορικής. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ειδικά και κλειστά συστήματα πληροφορικής. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια τα οποία ισχύουν σε εμά πέραν των πολιτικών και των πολιτικών κριτηρίων και αποφάσεων. Τώρα, γιατί δεν ενδιαφέρονται περισσότερε χώρε να προσχωρήσουν σε εμά. Δεν το Ακόμα δεν έχουμε διαφημίσει την EATC. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται ενδελεχώς οι στόχοι μας, το καταστατικό μας, ε, τότε όταν συζητούσαμε τη δημιουργία της EITC δεν είχαμε συζητήσει τη διεύρυνση. Είχαμε πει ότι εν ευθέτω χρόνο θα γίνει και η διεύρυνση. Ε, και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα έχουμε νέες χώρες που θα έχουν προσχωρήσει και δει το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο έχει μια πολύ ε, εμείς έχουμε μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση και πιστεύω ότι θα πείσουμε πολλές άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αξιωματούχο σύνδεσμο στη Ισπανό για την Ισπανία, ο οποίος ε, προετοιμάζει το έδαφος στην Ισπανία και καταγράφει τη στάση, την προσέγγιση της Ισπανίας. Είμαστε λοιπόν φρέσκοι, καινούργοι και τώρα αρχίζουμε την να διαφεμιζόμαστε την προβολή μας. Για τα αεροσκάφη, το στόλο, είμαι πολύ ικανοποιημένο για το μέγεθος του στόλου που έχουμε κάτω από επιχειρησιακό έλεγχο. Οι στρατιωτικές αερομεταφορές, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ ακριβές και πρέπει να βρούμε φθηνούς τρόπους μεταφοράς. Ε, γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιούμε, ε, ε, χρησιμοποιούμε την αρχή της υπεργολαβίας. Αναθέτουμε δηλαδή σε τρίτους ορισμένες μεταφορές. Και ο αρμόδιος για την ανάθεση σε εξωτερική ιδιωτικούς φορείς διαφόρων επιχειρήσεων κάθεται 100 μέτρα από το γραφείο μου. Ε, πρέπει να έχουμε μία ε, ε, προσέγγιση ανοιχτή, ε, να χρησιμοποιούμε κάθε δυνατό τρόπο συνεργασίας με τρίτους συνεργάτες. Υποστηρίζουμε Επίσης την παροχή ωφελών στα διάφορα πληρώματα, ε, την παροχή τεχνικής κατάρτισης, ε, τεχνικής εκπαίδευσης. Ε, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη στην Ευρώπη της βέλτιστης κατάρτισης εκπαίδευσης του προσωπικού αερομεταφορών και τώρα πηγαίνουν στη σχολή του Σαν Τζόζεφ στις Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίοι είναι πανάκριβοι, οι οποίοι είναι εξαιρετικά καλοί και επαγγελματικοί, για να εκπαιδευτούν. Και ακόμα ε, και η αμερικανική ε, αεροπορία, πολεμική αεροπορία ενδιαφέρεται για το πώς μπορεί να εμπλουτίσει το πρόγραμμά της, ας πούμε, με, ευρωπαϊκές, με ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Υποστηρίζουμε την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Θα διοργανώσουμε με ένα μεγάλο συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση μου έστειλε μια, μια πολύ ωραία επιστολή εξέτοντας αυτά τα θέματα και επίσης θα προεδρεύσω εγώ μία συνάντηση στη Σαραγκώσα για την κατάρτιση των στελεχών μας και θα προσπαθήσω να συμβάλλω όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να επανασχεδιάσουμε όλη αυτή την εκστρατεία επιμόρφωσης. Γιατί δεν περάσαμε μέσω του ΝΑΤΟ και ε, τη στρατιωτική ενσωμάτωση. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για επίπεδο διοίκησης. Εμείς είμαστε μέρος της στρατιωτικής δομής των τεσσάρων κρατών και αυτό είναι σημαντικό. Εγώ υποστηρίζω τους, το γαλλικό στρατό, τις γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις και θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Δεν ήταν λοιπόν επιχείρηση αυτή, επιχείρημα μάλλον εντός του, ΜΑΤΟ, του ΝΑΤΟ, προς ενσωμάτωση εντός του ΝΑΤΟ, ήταν μια ξεχωριστή διοικητική δομή η AATC. Um, Ευχαριστώ. Μία σύντομη ερώτηση. Για ποια συνθήκη μιλάτε, τη συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μία ε, σύμβαση με τον ΝΑΤΟ, γιατί μιλάτε για το 2012 και δεν κατάλαβα για ποια συνθήκη μιλάτε. Ναι, όχι, είναι η σύμβαση αυτών των τεσσάρων κρατών. Αυτό εννοούσα, δηλαδή προσδιορίζουν τη θέση που θα καταλάβει η Ευρωπαϊκή Διοίκηση Αερομεταφορών στα πλαίσια των εθνικών του πόρων. Πρέπει να προσέχω πάρα πολύ τι λέω γιατί ε, ο όρος ε, σύμβαση στα πλαίσια των διεθνών οργανώσεων είναι νομικά δεσμευτικός και άρα πρέπει να προσέχω ε, τι λέω. Πολύ ωραία στρατηγέ μου. Νομίζω ήσασταν σαφέστατος προς ικανοποίηση των συναδέλφων και του υποφαινομένου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη και για τις διευκρινήσεις σας. Όπως είπε ο Αντιπρόεδρος Λίζεκ, πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, διότι απηχεί αυτή τη νέα φιλοσοφία, δηλαδή ε, προσπαθούμε να πείσουμε τα κράτη να συνεργαστούν όχι μόνο στο, στρατιωτικό τομέα, στον τομέα των ενόπλων mm. δυνάμεων, αλλά και γενικότερα και ελπίζω να ε, διευρυνθεί ε, αυτή η δομή και να καλύψει και άλλους τομείς. Ε, πλέξατε το εγκόμιο τόσο πολύ της ε, διοίκησής σας στο Eindhoven, ε, οπότε ε, δεν ξέρουμε, μπορεί καμιά φορά να σας επισκεφτούμε όταν κάνουμε τέτοιες επιχειρήσεις στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας να σας να απευθυνθούμε σε εσάς να προσφύγουμε σε εσά. Τέλο πάντων ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια και θα είμαστε σε επαφή για να παρακολουθήσουμε ε, την εξέλιξη αυτή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και για να την επισκεφθούμε.